<coughs> Καλημέρα σε όλους. Αρχίζουμε τις ψηφοφορίες μας. Πρέπει να σας πω ευθύς αμέσως ότι δεν έχουμε διερμηνία προς τα βουλγάρικα. Πάμε στο πρώτο σημείο. Τη ημερήσιας διάταξη, απαλλαγή 2009 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν ε, ψηφίσουμε, έχει το λόγο ο εισηγητής ο κύριος Ήταλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, έχουμε ήδη διανύμει τον ε, κατάλογο πρόεδρε. Δεν θα έλθω σε λεπτομέρειε. Θα ήθελα όμω ω σκιώδη συγητή να εκφράσω τι ευχαριστίε μου, διότι ήταν εξαίρετη η συνεργασία και η βούληση για ε, συμβασμού. Πλευράς, για συμβασμό πλευράς του συγητή. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πολύ καλό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη υπόθεση. Για τα σημεία, για το σημείο 65, Και στο 506 έχουμε ένα μείον στο πρόσημο, πρέπει να διορθωθεί. Είναι συν. Ίσως να είναι αυτό ε, λάθος μόνο στο δικό μου αντίτυπο, αλλά ας διορθωθεί παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Αν είστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία και αφορά στην απαλλαγή 2009 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Η ψηφοφορία ξεκινάει. Προφορική τροπολογία είναι το πρωτότυπο. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 4, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παρακαλώ. Λοιπόν, διαδικαστικό. Εγώ νομίζω ότι η τέσσερα του κυρίου Αντρίσεν έχει... Α, ανάποδα, ανάποδα ήταν, εγκρίθηκε. Α, και το τρία της κυρίας Χέρτζοκ. Η πέντε πέρασε και η τρία έχει καταπέσει. Οχτώ. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 11. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 10. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 24. 24 24 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 27 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 29 υπέρ πέρας κατά απορρίπτεται συγγνώμη 28 αρχίζει ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 39 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. 31 χωριστά. Στο πρώτο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έχουμε έναν παραπανήσιο για το ΕΛΚ. Ένας παραπάνω ψήφισε για το ΕΛΚ. Απορρίπτεται. 32 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τριάν No, no, questo. Ok, 35. Emendamento 35, la votazione aperta. 35 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας Ok, Okay. Votazione chiusa. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 34 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 37 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 38 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 39 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 41 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 42 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 44 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας απορρίπτεται. 46 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας απορρίπτεται. 45, όχι, όχι, 48. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 47 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 49 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 50 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 51 αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας. Ένας παραπάνω πάλι. Εγκρίνεται. 53. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 57 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 58 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 59 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 60. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 61. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 62. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 63 αρχίζει η ψηφοφορία πέρασε εγκρίνεται 64 άρχεται η ψηφοφορία Εξήντα έξι αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε απορρίπτεται 67 αρχίζει η ψηφοφορία πέρασε απορρίπτεται 68 αρχίζει η ψηφοφορία πέρασε εγκρίνεται 69 αρχίζει η ψηφοφορία Πέρασε. Εγκρίνεται. 70. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 71. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 72 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 73 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 74 αρχίζει η ψηφοφορία πέρασε εγκρίνεται 75 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 76 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 77 σε δύο, μέρη, δύο τμήματα. Πέρας ψηφοφορίας για το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 78. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 79. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 80 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 81 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 82 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 83 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 84 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 85 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 86 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 87 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 88 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 89. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 90. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 91. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασα. εγκρίνεται 92 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 93 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 94 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 95 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 96 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 97 αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 98 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 99. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 100 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 101 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 102 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 103 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 105 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 106. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 104 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 108 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται η 110 αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 112 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 109 αρχίζει, συγγνώμη, 111 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 113. Αρχίζει η ψηφοφορία. Όχι, όχι. Α, η 115 τότε. 115 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 116 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 114 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 118 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 119 αρχίζει ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θα ήθελα να προτείνω μια προφορική τροπολογία για την 120 τροπολογία το IN 2011 να γίνει after 2011, δηλαδή επιμένει να υπάρξει διακοπή μετά το 2011. Ξέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει η έχει ξεκινήσει η προπαρασκευή, άρα νομίζω ότι στόχος μας δεν είναι το παρελθόν, αλλά το μέλλον. Όχι in 2011, after, όχι κατά το, μετά. Ωραία, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει να ψηφίσουμε την 120 με την προφορική τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 121. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 122. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 123. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 124. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 126. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 125. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 128 αρχίζει η ψηφοφορία πέρασε εγκρίνεται 127 αρχίζει η ψηφοφορία πέρασε ψηφοφορία εγκρίνεται 129 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται 131 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 130 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 132 αρχίζει η ψηφοφορία τελειώνει η ψηφοφορία εγκρίνεται 133 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 134 αρχίζει η ψηφοφορία τέλος απορρίπτεται 135 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 136 αρχίζει. Τέλος. Απορρίπτεται. 137 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 138 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 139 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 140. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 143. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 141 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 144 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 145. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να μου δώσετε το λόγο όταν θα έχουμε ψηφίσει την 147 μετά από την 147. Μετά την ψηφοφορία της 147 σας ευχαριστώ. Τροπολογία 145 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 146 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 147 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται παρακαλώ συνάδελφε Ματίο ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εγώ είμαι κατά της προφορικής τροπολογίας αυτό είναι ένα και δεύτερο θέλω να ψηφίσουμε την τροπολογία 150 του κυρίου Οντί και δική μου πριν από την 148. Δεν καταλαβαίνω γιατί την τροπολογία μου 150 την ψηφίζουμε μετά την τροπολογία 148. Διότι η τροπολογία μας θυμίζει, ε, ε, υπενθυμίζει τους όρους της συνθήκης για τους τρεις τόπους εργασίας. Μα τον κατάλογο ψηφοφορίας ε, τον ετοίμασε η γραμματεία και πρέπει να συνεχίσουμε κατά, με αυτή τη σειρά. Εκτός και αν όλοι συμφωνείτε να το αλλάξουμε. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν τον κατάλογο ψηφοφορίας. Να μου εξηγήσετε όμως γιατί. Γιατί μία τροπολογία που κάνει υπόμνηση, στην, που αναφέρεται στη συνθήκη, και μου το βάζετε μετά το 148. Μα είναι πραγματικά κατανόητο, Αλλά εξηγήστε το μου με επιχειρήματα. Η εξήγηση είναι η εξή. Ο κανόνας λέει ότι πρέπει να ψηφίζουμε πρώτα το κείμενο το οποίο πάει μακρύτερα από το κείμενο. Η τροπολογία της κυρίας Σαλνεμούζε πάει πιο μακριά από τη δική σας τροπολογία. Έχετε όμως δίκιο, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε την τροπολογία σας μετά την τροπολογία της κυρίας Σαλντεμόζε, έστω και αν ψηφιστεί η τροπολογία Σαλντεμόζε, διότι είναι συμβατή η δική σας. Και φυσικά σημειώσαμε όσα είπατε για την προφορική τροπολογία, την οποία δεν θα ψηφίσουμε. Allora, votiamo eh, l'emendamento orale. Θα ψηφίσουμε τώρα την προφορική τροπολογία χωριστά. Λοιπόν, πρώτο τμήμα. Όχι, λέει η γραμματεία. Α. Il paragrafo 99, sì. Παράγραφο 99. Την παράγραφο 99 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Approvato. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 148. Αρχίζει η ψηφοφορία. Όχι! Όχι, φωνάζει η κυρία Ματιέ. Μα δεν έπρεπε να ψηφίσουμε για την προφορική τροπολογία, διότι εγώ έφερα αντιρρήσεις. Αλλά γιατί. 148, σαραντοχτώ. Η κυρία Γκρέσλε. Ε, μα τι ψηφίζουμε τέλος πάντων. Είπαμε η 148 το πάει μακρύτερα από την 150. Γι' αυτό ψηφίζουμε καταρχήν την 148 και μετά την 150. Μα δεν αλλάζει ο συσχετισμός. Μα, μας είπατε πριν από μερικά λεπτά ότι θα ψηφίσετε πρώτα την 150 και μετά την 148. Μα η 150 τροποποιεί περισσότερο το άρθρο από ότι... Κύριε Γκρέσλε, το πιστεύετε, δεν ξέρω, πάντως ο πρόεδρος μου δώσει το λόγο, αν μου επιτρέπετε λοιπόν. Η τελευταία ψηφοφορία έφερε, αφορούσε την 147. Και βλέπω στον κατάλογο το δικό μου ότι προβλέπεται χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 99. Και παρακαλώ να μην το ξεχάσουμε. Η ψηφοφορία Έγινε μεν, αλλά δεν ανακοινώθηκε αποτέλεσμα. Μπορείτε παρακαλώ να μας ενημερώσετε για το αποτέλεσμα του σχετικό με την παράγραφο 99. Ποια ήταν η έκβαση της ψηφοφορίας. Θέλω να ξέρω ποια ήταν η αναλογία ψήφων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Θέλω απλώς να επισημάνω ότι το ζήτημα του Στρασβούργου μπορεί να προξενήσει συνθήκες εμφυλίου πολέμου μέσα στις ομάδες. Γι' αυτό θέλουμε να ξέρουμε ποιες ήταν οι αναλογίες της ψηφοφορίας. Λοιπόν, ψηφίσαμε την παράγραφο 99 και υπερψηφίστηκε η 99, το είπαμε και πριν. Η παράγραφος 99 και ψηφίζαμε την 148. Θέλω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Πόσοι υπέρ, πόσοι κατά σας εκλήπαρο, δώστε μου το αποτέλεσμα. Ωραία να ξαναψηφίσουμε. Ξαναψηφίζουμε την παράγραφο 99. Ε, και αν αλλάξει η ψηφοφορία, φωνάζει ο κύριος Ριβελίνη χωρίς μικρόφωνο, Ο πρόεδρος πρέπει να αποφασίσει, ο πρόεδρος πρέπει να αποφασίσει. λοιπόν, να το ξαναψηφίσουμε. Allora. Allora. Λοιπόν, να σα πω, να σας πω. 27 ψηφίσαντες, 18 υπέρ, 9 κατά και καμία αποχή. Ούτως εψηφίστη 99. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα ψηφίσουμε την 148 ή την 150. Αυτή ήταν η αμφιβολία μας. Πρόεδρε, τον κατάλογο. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να τροποποιηθεί το αποτέλεσμα και να προξενηθεί σύγχυση. Παρακαλώ να ακολουθήσουμε όπως έχουμε τη σειρά μας τον κατάλογο. Εγώ προσωπικά έδωσα το λόγο σε όλους. Ο κατάλογος λοιπόν ψηφοφορίες δεν θα πρέπει να αλλάξει. Κύριε Πρόεδρε, όποια και να είναι η σειρά, 148 ή 150, συμφωνούμε σε αυτό που διευκρίνησε η Γραμματεία. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ψηφίσετε την 148 πριν από την 150, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα θα ψηφιστεί η 150 μετά. Άσχετα δηλαδή από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Βεβαίω να ψηφίσουμε λοιπόν την 148 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται η 148. 150 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 151 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 152 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 153 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 154 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 155 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 156 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 157 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται 159 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 160 αρχίζει Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 161 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται. Η τελική απόφαση αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τελικό ψήφισμα αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τέλεια. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Abbiamo adesso eh, il discarico. Chiedo Απαλλαγή για τα άλλα θεσμικά όργανα. Η συγητής είναι ο κύριος Ριβελίνη. Θέλει το λόγο ο κύριος Ριβελίνη. Μόνο για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεργασία, ένα δύσκολο ντοσιέ. Πιστεύω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά, πήρα το λόγο μόνο για να ευχαριστήσω, το ξαναλέω. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Ψηφίζουμε την απαλλαγή 2008 λέει ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Τροπολογία 1 αρχίζει ψηφοφορία. La votazione Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική απόφαση. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική απόφαση, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Okay. Questo qua, Corte di Giustizia.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 Τροπολογία 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 6. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Τροπολογία 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 9. Ε, ναι, χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 για την παράγραφο 8 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 13. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Κυρία Αγιάλα. Αποσύρω την 16 την τροπολογία μου υπέρ της 17 του κυρίου Ριβελίνη. Ψηφίζουμε την 17, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε αμπλόκ τις τροπολογίες 23-33. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνονται. 21. Αρχίζει η ψηφοφορία. Όχι, όχι, όχι. Διορθώνει το πρόεδρος. 22. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 32 αρχής ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Πρόεδρε θα ήθελα να προτείνω στην κυρία Μακοβέη χωριστή ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα να ψηφίσουμε χωριστά μέχρι την πρώτη τελεία και μετά από εκεί που λέει επίσης και σε επίπεδο της Ένωσης. Και τονίζει ότι θα έπρεπε να είχαμε δυνατότητες εξοικονόμησης κλπ. Και θα καταψηφίσει η ομάδα μου και το δεύτερο τμήμα φαντάζομαι ότι και ο κύριος Σοντή θα πρέπει να το καταψηφίσει. Γιατί πάλι παίζει στο Στρασβούργο εκεί, λέει η κυρία Γιάλα. Λοιπόν, 34 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Μα το δεύτερο τμήμα είναι Στρασβούργο, λέει η κυρία Γιάλα. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα όπως ε, τροποποιήθηκε. Παρακαλώ. Εγώ πρόεδρε θα ήθελα να το πω δημόσια. Εσείς κάποια στιγμή μιλήσατε για μια προφορική τροπολογία που δεν την έχουμε στον κατάλογο ψηφοφορίας και φαντάζομαι ότι ήταν η προφορική τροπολογία της κυρίας Γκρέσλε στην οποία δεν επανήλθαμε. Εγώ θα ήθελα διότι είχαμε μια δική μου τροπολογία και μετά εξαφανίστηκε η 12. Στην παράγραφο 8, ποια ήταν αυτή. Α, δεν ήταν η δική μου, δεν είναι η δικιά μου. Α, δεν ήταν η δικιά μας αυτή. Ψηφίσαμε, ψηφίσαμε για την 8 προφορική τροπολογία. Το καταλαβαίνω, αλλά Θέλω να το καταγράψετε επειδή δεν το είχα στο δικό μου κατάλογο ψηφοφορίας ότι ήμουνα κατά... Το ψηφίσατε. Ναι, ναι, μα ασυνείδητα το ψηφίσαμε, λέει η κυρία Γιάλα. Εγώ ήμουνα κατά και να το γράψετε και καθαρά και εξάστερα στα πρακτικά ότι ήμουνα κατά. Αλλά μπερδεύτηκα. Χωρίς μικρόφωνο. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, αλλά να μπει στα πρακτικά, να μπει στα πρακτικά. Μα ήσασταν σαφέστατοι. Θέλει η κυρία Γιάλα Σέντερ να καταγραφεί στα πρακτικά η ψήφο τη. Ωραία. Πάμε. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό που είπε Δεν έδωσα κανένα μήνυμα εκ τη ομάδα μου προ το παρόν, διότι η προφορική τροπολογία στην οποία αναφέρεστε δεν προβλεπόταν στον κατάλογο και ως εκ τούτου η θέση της ομάδος μου θα ήταν μάλλον αρνητική επάνω στην προφορική τροπολογία. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Ωραία, σημειώνουμε και τα του κυρίου Γκάγερ. Ψηφίζουμε το τελικό ψήφισμα, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται τελειώσαμε με το Συμβούλιο Passiamo adesso alla votazione. Πάμε στην ψηφοφορία για την απαλλαγή 2008 του δικαστηρίου. Ψηφίζουμε το σχέδιο απόφασης, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και μετά ψηφίζουμε το ψήφισμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τώρα, απαλλαγή 2009 του ελεγκτικού συνεδρίου αρχίζει η ψηφοφορία για την πρόταση απόφαση πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τις τροπολογίες. Ένα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δύο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Συμβιβασμός 2. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τελικό ψήφισμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Passiamo adesso alla votazione per il discarico 2009. Απαλλαγή 2009 για την ΟΚΕ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Παρακαλώ. Λέει ο κύριος Ριβελίνη, υπάρχει μία προφορική τροπολογία ή δυνατόν να τη διαβάσουμε. Επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Η τροπολογία λέει, έχει τη γνώμη ότι είναι λογικό να αναβληθεί η απαλλαγή για την ΟΚΕ εν αναμονή των συμπερασμάτων της έρευνας της Όλαφ. Να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία του κυρίου Ριβελίν. Θέλετε να την, Θέλετε να την επαναλάβω. Ωραία. Έχει τη γνώμη ότι είναι λογικό να αναβάλουμε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΟΚΕ αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από τον έλεγχο της ΟΛΑΦ. Έχετε αντιρρήσεις? Όχι, όχι. Να ψηφίσουμε τότε την προφορική τροπολογία του κυρίου Ριβελίνη. Αρχίζει η ψηφοφορία.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 13 ναι. κατά, 12 υπέρ, αποφάσισαν την αναβολή της απαλλαγής. Και σε ένα βαθμό μπαίνουν τα κείμενα αυτά και στις ε, τροπολογίες του εισηγητή, δηλαδή τα λέμε δύο φορές. Ας περιπτώσει, δεν περιμέναμε ότι θα γίνει αυτό. Και θέλω να πω ότι νομοτεχνικά καλό θα ήταν να κοιτάξουμε να τα προσαρμόσουμε για να μην έχουμε εσωτερικές αντιφάσεις. Έτσι. Ευχαριστώ. Eh, Εσείς λέτε ότι στην τροπολογία 2 τη συναδέλφου Σέντερ ήδη συμπεριλαμβάνονται τα περιεχόμενα της προφορικής τροπολογίας του κυρίου Ριβελίνη. Να ψηφίσουμε την τροπολογία 2. Αυτό λέτε αν κατάλαβα καλά. η προφορική σας τροπολογία θα έμπαινε στο δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 2. Μα η προφορική μου τροπολογία διευκρινίζει, εμβαθύνει. Σίγουρα συνεισφέρει στη συζήτηση, βοηθάει. Διότι διευκρινίζει την τροπολογία 1 της κυρίας Αγιάλα. Εγώ για το 2, για το 2 λέω. Όχι, σε σχέση με την τροπολογία 1 της κυρίας Αγιάλα, το δεύτερο τμήμα. Η τροπολογία 1 που εγκρίθηκε της κυρίας Αγιάλα. Έχουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας μου που ψηφίσαμε. Στην τροπολογία 1 το ψηφίσαμε αυτό. Presidente, noi abbiamo, approva- noi abbiamo sì, sì, no, approvato chiaro, solo l'emendamento 1. Εμείς εγκρίναμε την τροπολογία 1. Il problema è che noi abbiamo votato l'emendamento 1 e poi abbiamo votato... Το πρόβλημα είναι ότι ψηφίσαμε την τροπολογία 1 και μετά ψηφίσαμε το ψήφισμα. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 2 που παρουσίασε η κυρία Γιάδα. Το δικό μου δύο δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης πλέον διότι πρέπει να ψηφίσουμε την 9α που είναι το δεύτερο τμήμα της προφορικής τροπολογίας που αντικαθιστά το σκεπτικό το οποίο φαίνεται τώρα ως βίο αλλά έχει πλέον ξεπεραστεί διότι πρέπει να βάλουμε το δεύτερο τμήμα της προφορικής τροπολογίας που είναι το 9α. Οι προφορικές τροπολογίες του κυρίου Ριβελίνη πλέον δεν έχουν νόημα διότι έχουμε να ψηφίσουμε τώρα το δεύτερο τμήμα της δικής μου τροπολογίας. Αλλά δεν ξέρω πού είναι ο κατάλογος, ο πραγματικός κατάλογος της ψηφοφορίας. Μου φαίνεται σαφές αυτό το οποίο λέει η κυρία Γιάλα. Ψηφίσαμε την τροπολογία 1, ψηφίσαμε και το ψήφισμα και η κυρία Γιάλα λέει ότι μόνο το δεύτερο τμήμα της προφορικής αστροπολογίας πλέον υφίσταται.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 Eh, Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία αριθμός δύο της συναδέλφου Αγιάλα. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα και δεύτερο τμήμα. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 2 της κυρίας Σέντερ αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 2 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψυχοφορίας. Εγκρίνεται. Η προφορική τροπολογία σε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία D η Δέλτα. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ε, προφορική τροπολογία ε, αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σίγμα ταφ, F, λατινικό, αρχής ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός ένα, αρχίζει. Ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία ή Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Προφορική τροπολογία J, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίες, Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα ούτως τροποποιημένο, αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίες. Τελικό ψήφισμα. Τώρα. Απαλλαγή 2009 της Επιτροπής των Περιφερειών. Αρχίζει η ψηφοφορία για το σχέδιο απόφασης. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τον συμβιβασμό 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα ούτως τροποποιημένο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Απαλλαγή 2009 Ευρωπαίος διαμεσολαβητής. Σχέδιο απόφασης. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελικό ψήφισμα, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Απαλλαγή 2009 Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων αρχίζει η ψηφοφορία για το σχέδιο απόφασης πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται ψηφίζουμε το τελικό ψήφισμα, αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Ριβελίνη για τη δουλειά του. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου η αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βασική εκπαίδευση στην υποσαχάρη Αφρική και την Ανατολική Ασία. Ο συνάδελφος Στάις έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως καλό θα ήταν καταρχάς να ε, μιλήσει το ελεγκτικό συνέδριο που μας διαβίβασε και το εξαιρετικό αυτό έγγραφο. Θα ήθελα να ακούσω πρώτα το ελεγκτικό συνέδριο, να συνοψίσει τη δουλειά του και μετά εγώ θα σχολιάσω εφόσον είναι απαραίτητο. Συμφωνείτε? Σύμφωνο. Ο κύριος Κίστ του ελεγκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον εισηγητή σας κύριο Στάς για την ενδελεχή και εξαιρετική ανάλυση της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου όπως αυτή παρουσιάζεται στο έγγραφο εργασίας του. Η βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι σημαντικός παράγοντας καταπολέμησης της φτώχειας. Αυτό κατοπτρίζεται στην ε, κίνηση ΕΦΑ, ε, παιδεία για όλους, καθώς και στους αναπτυξιακούς στόχους ε, της χιλιετίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αναλάβει πρωτοβουλίε ε, με, με ειδικού στόχου ε, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που θα πρέπει να παρέχεται σε όλα τα παιδιά, την κατάργηση διαφορών ε, λόγω στην παροχή τη εκπαίδευση και γενικώ στη βελτίωση τη παιδιάς τη ποιότητα παιδεία. Έχουμε λοιπόν αυτού του τρει-τέσσερι βασικού στόχου και θα πρέπει να του αξιολογήσουμε, να δούμε κατά πόσον συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την ε, βελτίωση της εκπαίδευσης και κατά πόσον δεύτερον η Κομισιόν διαχειρίζεται τις παρεμβάσεις στον τομέα της ε, παιδείας με το σωστό τρόπο. Εμείς επικεντρώσαμε ε, την προσοχή μας σε διάφορες περιοχές ποσαχάρια Αφρικής και της Νοτελικής Ασίας, σε υποπεριοχές συγκεκριμένα όπου υπήρχαν πιο έντονα προβλήματα στον τομέα της εκπαίδευσης. Πριν σας ενημερώσω για τις κυριότερες παρατηρήσεις του ελληνικού Συνεδρίου, πρέπει να σας πω ότι η ανάπτυξη εκπαίδευση στο μεγαλύτερο τμήμα τη γίνεται στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων τα οποία ε, τα αναλαμβάνουν οι ε, κυβερνήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει άμεση εξουσία για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Είναι σημαντικό λοιπόν για την Κομισιό να θεσπίσει σαφή και ρεαλιστικούς δείκτες και στόχους ε, για τη διατήρηση ενός πραγματικού διαλόγου με τις κυβερνήσεις, εταίρους και άλλους φορείς. Και αυτό βέβαια ισχύει για οποιαδήποτε αναπτυξιακή ε, βοήθεια. Έχοντας αυτό υπόψη λοιπόν, κοιτάζουμε τώρα τα συνολικά αποτελέσματα των ε, ελεγχθέντων προγραμμάτων και την τομεακή υποστήριξη ε, όπου είδαμε το 45% των αποτελεσμάτων ε, των δικτών επιτέφεσαν και έχουμε και κατά 30% πρόοδο. Σε ό,τι αφορά τα ελεγχθέντα προγράμματα, σε περισσότερες περιπτώσεις απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αλλά είχαν, ήταν μικρής κλίμακας. Υπήρξαν επίσης βελτιώσεις σε διάφορες χώρες για την εξασφάλιση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για, όλους, για όλα τα παιδιά. Είναι όμως γενικά βραδία η πρόοδος. Θα πρέπει ε, να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες, ιδίως για την ολοκλήρωση του πλήρους κύκλου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί αυτό δεν επιτυγχάνεται, ε, πολλό μάλλον, ε, πόρο απέχει, μάλιστα σε πολλές από τις φτωχότερες χώρες. Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των διαφορών λόγω γίνονται προσπάθειες, τα στοιχεία όμως ε, νομίζω ότι συγκαλύπτουν ακόμη τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ διαφόρων κοινωνικών και περιφερειακών ομάδων. Η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης επίσης εξακολουθεί να είναι ζήτημα και παραμένει βασικότερη πρόκληση. Πολύ λίγες από τις αναμενόμενες πρόοδες έχουν επιτευχθεί. Το, το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι η προτεραιότητα που δίνεται ε, στις, ε, στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας που είναι ένα ποσοτικοποιημένο εργαλείο θα βοηθήσει στην ε, ανάπτυξη της ποιότητας εκπαίδευσης. Πάντως ε, δείχνουν όλα αυτά μόνο μια μερική πρόοδο. Δεν θα πρέπει βέβαια να υποτιμήσουμε τα επιτεύγματα. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν αδυναμίες και δεν μπορούμε να τις καταλογίσουμε μόνο στην κοινότητα των δωρητών ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων, τον προγραμματισμό, υπήρξαν κάποια προβλήματα που εν μέρει επηρέασαν την παράδοση των αποτελεσμάτων. Στην έκθεση εκτίθενται αναλυτικά όλα τα στοιχεία και βέβαια συνοδεύεται η έκθεση αυτή και από τι συστάσει του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν μια ευρία, ένα ευρύ ε, φάσμα μεθόδων, πρέπει να τις συνδυάσουμε σε αυτές τις μεθόδους ε, για να ε, στηρίξουμε τις προσπάθειες αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται από μη κρατικού φορείς. Και θα πρέπει να στοχεύσουμε ιδίω σε παιδιά τα οποία είναι δύσκολο να τα προσεγγίσουμε. Έχουμε διάφορους στόχους. Έχουμε τη μέθοδο ε, της στήριξης μέσω του γενικού προϋπολογισμού που είναι το βασικό εργαλείο θα πρέπει να υπάρξει και εμπειρογνωμοσύνη. Οι δείκτες επιδόσεων θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στη συστηματική παρακολούθηση και αναθεώρηση και στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Υπάρχουν κάποια βασικά μηνύματα ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου, τα έχετε στην έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες της Κομισιόν για την πολύ επικοδομητική τους συνεργασία σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, συνάδελφο Στάς. Ehm, eh, σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το ελεγκτικό συνέδριο. Όπως προείπα, εργάστηκε εξαιρετικά. Η ειδική αυτή έκθεση εγκύπτει και στο γενικότερο ζήτημα της χρηματοοικονομικής βοήθειας. Είναι ένα επίκαιρο θέμα αυτό. Πρώτον, διότι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού έχουμε εξετάσει αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο της απαλλαγής του Ταμείου Ανάπτυξη, αλλά και για την πράσινη βίβλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση αναφέρεται ε, στη δημοσιονομική στήριξη, στη στήριξη μέσω του προπολογισμού. Θα ψηφίσουμε μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή μα την επόμενη εβδομάδα, μια γνωμοδότηση που τα απευθύνουμε προ ε, την Επιτροπή Αναπτυξιακή ε, Βοήθεια. Είναι πολύ λοιπόν εύστοχη έκθεση, επίκαιρη, αναφέρει κενά, αλλά και αποτελέσματα τα οποία επιτεύξαν παρά τα κενά που υπάρχουν. Και έχουμε και κάποια στοιχεία. 45% των δικτών έχουμε επιτυχία εκεί και η Κομισιόν λέει ότι εκτός αυτού, εκτός αυτού του στοιχείου το 30% των δικτών δείχνουν σημαντικά ε, σημάδια βελτίωση. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου και νομίζω βέβαια ότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε στις δάφνες αυτές, αλλά θα πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι η εκπαίδευση, η παιδεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κομβικό, αν θέλετε, υπόστρωμα και τα κονδύλια τα οποία ε, εμείς διαθέτουμε για την εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν πραγματικά αποτελέσματα και να ωφελούν τους πολίτες. Γι' αυτό στις συστάσεις μας ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν είναι δυνατό να μας κάνει μία επισκόπηση κατανεμημένη αναχώρα, ε, να δούμε τα ποσά αναχώρα και το εύρος, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στο έργο του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό το οποίο είναι λίγο περίεργο και το λέω για νιωστή φορά και σε σχέση με την ιωστή έκθεση αυτή του ελεγκτικού συνεδρίου. Γίνεται αναφορά στι ελλείψει, ελλείψει εξειδικευμένου προσωπικού. Εγώ ξέρω ότι είναι λεπτό το ζήτημα του προπολογισμού. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με την ανακύκλωση και την αναλλαγή του προσωπικού. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλοι γνωρίζουμε ότι οι προσπάθειες που γίνονται στον τομέα της εκπαίδευσης είναι σημαντικές για το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όταν διαπιστώνουμε ότι ορισμένες αντιπροσωπείες της Κομισιόν δεν έχουν το επαρκές προσωπικό από πλευράς προσόντων και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα βοήθειας για την εκπαίδευση. Εκεί έχουμε προβλήματα. Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να σκεφτούμε στο Κοινοβούλιο πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την αρμόδια Επιτροπή για την ε, Αναπτυξιακή Συνεργασία, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Προπολογισμών. Όλε αυτέ τι αρμόδιε επιτροπέ. Και θα πρέπει επίση να δούμε πώ μπορούμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα τη μη επαρκού στελέχωση των αντιπροσωπιών. Και σε ένα από τα επόμενα συμπεράσματά μου, στι επόμενε συστάσει μου, μου ζητώ κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην παραμείνει ένα κενό γράμμα. Να μην τη βάλουμε σε ένα σιρτάρι και αυτή την έκθεση για να πιάνει σκόνη όπως όλες οι άλλες. Θα πρέπει αυτή την έκθεση να ε, την παρακολουθούμε, να της δώσουμε συνέχεια. Τέσσερα σημεία θέλω να σχολιάσω. Πρώτα απ' όλα, τι είναι σημαντικό, ποιότητα τη εκπαίδευση. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το λέει ρητά και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχει και ένα έγγραφο εργασία ε, του Φεβρουαρίου που λέει καλύτερη εκπαίδευση για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Είναι ένα έγγραφο το οποίο δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να χρησιμοποιούν αντιπροσωπείε. Αυτό το έγγραφο χρησιμεύει για την αξιολόγηση τη ποιότητα τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση. Εξού και ρωτώ την Εκτελεστική Επιτροπή ποια άλλα μέτρα και ποιε άλλε πρωτοβουλίε θα ή μπορεί να αναλάβει για να βελτιώσει την ποιότητα και την παρακολούθηση τη εκπαίδευση. Δεύτερο σημείο. Απάτη, διαφθορά. Ε, από ό,τι λέγεται ξεκάθαρα υπάρχουν περιπτώσεις απάτη σε διάφορες χώρες και κάποιες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι καθηγητές φαντάσματα, ε, δηλαδή εκτοπλάσματα. Καθηγητές που υπάρχουν μεν αλλά ε, δεν εμφανίζονται και δεν παραδίδουν κανένα μάθημα ιονοί καθηγητέ τέλο πάντων. Τι κάνουμε με, αυτούς, με αυτά τα κρούσματα, με αυτού του είδου την απάτη. Τρίτο σημείο. Εκτέλεση η εκτέλεση ενό προγράμματο χρειάζεται και στατιστικά στοιχεία, μια παρακολούθηση. Αυτό δεν γίνεται. Πώ θα το διορθώσετε, κύριε και κύριοι τη Κομισιόν, το έχετε σκεφτεί και τελευταία παρατήρηση. Η συμμετοχή των κοριτσιών και των ε, γυναικών. Πολύ χαμηλή είναι η συμμετοχή από ό,τι φαίνεται και το έχω σε επισημάνει και στην έκθεση της, ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αυτό σχετίζεται και με άλλες παραμέτρους, υποδομές, ε, υγιεινή. Και θέλω να δω ποια στοιχεία θα ε, τι θα κάνει η Επιτροπή για να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Οι σανψόμενες χώρες πρέπει και τα κορίτσια να έχουν τη βασική εκπαίδευση. Και πρέπει να πω ότι πολύ συχνά οι γυναίκες που έχουν αποφεληθεί από μια ποιοτική εκπαίδευση είναι αυτές οι οποίες τελικά αναλαμβάνουν ε, την ανάπτυξη στις χώρες τους και αναλαμβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες. Φαντάζομαι ότι μόλις δώσετε το λόγο στην Κομισιόν θα έχω όλες τις απαντήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριε Σιγητά και μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Δεν χρειάζεται να πω ότι αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση και για την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου και για την δουλειά που έχει κάνει ο σα. Τα αποτελέσματα που διεπιστώνουμε και ότι δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε με βέβαια αφνές μας, συμφωνώ σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Μιλούμε για 67% των στόχων που ήλιο υλοποιήθηκαν. 75% των στόχων που υλοποιήθηκαν. Και επίσης, <clears throat> θα ήθελα να επισημάνω ότι εμεί παρακολουθούμε και τις μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές των κρατών εταίρων σε θέματα εκπαίδευσης όπως και στις άλλες ε, πολιτικές, τομεί πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια οι αντιπροσωπείες μας, όπως και εμείς εδώ, να έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να αναλύουμε κατά τρόπο πολύ προσεκτικό και περιστατωμένο τις πολιτικές σχετικές με την εκπαίδευση των κρατών εταίρων με δείκτες βελτιωμένους, όχι μόνο για input αλλά και για αποτέλεσμα δείκτες που να εστιάζονται στην ποιότητα. Και η ποιότητα βέβαια είναι από τα πολύ σημαντικά στοιχεία. Γιατί θα οδηγήσει σε μια ουσιαστική βελτίωση, όχι μόνο στον, αριθμό των ε, παιδιών που θα πάρουν στο σχολείο, αλλά το τι θα κάνουν βγαίνοντας από το σχολείο. Δηλαδή τι θα μάθουν. Δείκτες ε, που θα είναι εστιασμένοι στην μάθηση θα είναι κατάλληλοι για την προσμέτρηση αυτών των αποτελεσμάτων. Η ποιότητα, θα πω επίση δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των διδασκόντων που ασχολούνται στον κλάδο. Εξαρτάται επίση και το είπατε κι εσείς, από την παρουσία τους στο σχολείο. Επομένως, οι συχνές απουσίες είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Αν και πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί αυτοί οι διδάσκοντες καθηγητές δεν εμφανίζονται στο σχολείο, γιατί είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά απουσίας. Γιατί, διότι φερειπίν μερικές φορές χρειάζονται συμπληρωματικό εισόδημα και έτσι απασχολούνται κάπου αλλού. Ή άλλοτε, για λόγους άσχετους, γιατί η φερειπίν χρειάζεται να πάνε επί τόπου να πληρωθούν σε κάποιο ταμείο, όπως στην, ε, στον Ήγηρε παραδείγματι. 15 μέρες το χρόνο υπάρχει απουσία δασκάλων από τα σχολεία, διότι πρέπει να πάνε στην αρμόδια υπηρεσία να πληρωθούν. Άρα χρειάζονται και καινοτόμε λύσει, να βρούμε λύσει διαφορετικέ για το πώ θα καταβάλει το μισθό σε αυτών των δασκόντων. Έγινε λόγο ε, για χρήση του ε, κινητού τηλεφώνου, μέσω του κινητού τηλεφώνου να γίνονται πληρώμε. Εγώ δεν είμαι ειδική σε αυτέ τι νέε τεχνολογίε, αλλά πάντω υπάρχουν λύσει και μπορούμε να τις ε, ζητήσουμε. Έγινε λόγος λοιπόν για το φαινόμενο των συχνών απουσιών. Θα σας δώσω ένα πολύ ενδιαφέρον ε, παράδειγμα από την εμπειρία μας στη Μαδαγασκάρη, η οποία έκανε χαρτογράφηση αυτών των ε, εικονικών διδασκόντων τους προσέφερε αποζημίωση για να τους απομακρύνει από το σχολείο και να τους βγάλει από τη μισθοδοσία και παρά τις αποζημιώσεις αυτές φαίνεται ότι έχουν δημοσιονομικά κάποια ωφέλη ε, στη Μαδαγασκάρη, διότι παρά το ότι κράτησε αρκετό καιρό αυτή η χαρτογράφηση, μπορούσαν να εξοικονομήσουν πόρου. Άρα χρειάζεται η βούληση από πλευρά τη κυβέρνηση, χρειάζεται η παρακολούθηση, αλλά βέβαια χρειάζεται και η σύμπραξη όλων των ε, παραγόντων του τομέα. Και επίση θα ήθελα να υπογραμμίσω άλλο ένα ζήτημα που είναι αυτό τη διακυβέρνηση. Όσο αφορά εμά, εδώ έχουμε να κάνουμε με το ζήτημα του domestic accountability, δηλαδή τη λογοδοσία σε τοπικό επίπεδο. Πολλέ είναι οι πρωτοβουλίε που προλαμβάνονται στο θέμα αυτό, πώ δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια ή η κοινωνία των πολιτών ή το, το, τα τοπικά ελεγκτικά συνέδρια ούτω υπήν μπορούν να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι πόροι σε κάθε χώρα και σε κάθε τομέα. Και εδώ λοιπόν προσπαθούμε να ενισχύσουμε αυτή τη διάσταση και η δημοσιονομική στήριξη είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε ε, την κατάσταση. Επίσης αναφερθήκατε στο ζήτημα της ε, πρόσβασης στα σχολεία για τα κορίτσια. Για μας, ασφαλώς το γνωρίζετε, έχει τεράστια σημασία η, η συμμεταχείριση και σε αυτόν τον τομέα. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι πέραν πολιτισμικών ε, λόγων που μπορεί να επηρεάζουν ή και υγειονομικών, που όμως θα μπορούσαμε σχετικά εύκολα να επιλύσουμε, ε, μπορεί ο λόγος ε, για το ότι δεν πηγαίνουν τα κορίτσια στο σχολείο να είναι το ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες δασκάλες. Δηλαδή όταν έχουμε γυναίκα δασκάλα είναι πιο εύκολο να πάει το κορίτσι στο σχολείο. Το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό. Τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οθήσουμε και τις γυναίκες να αναπτύξουν δραστηριότητα ε, και στον ε, ε, και στο δευτεροβάθμιο βέβαια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο στην πρωτοβάθμια, για να μπορούν να παίξουν το ρόλο του διδάσκοντος στη συνέχεια και να ενισχύσουμε έτσι και την παρουσία των κοριτσιών στα σχολεία, πέραν βέβαια και του άλλου ζητήματος που είναι οι μεγάλες αποστάσεις από το σπίτι στο σχολείο ή του κινδύνου να υποστούν βία στο δρόμο, στη μετάβασή τους δηλαδή στο σχολείο. Όλα αυτά με οδηγούν στο εξή συμπέρασμα, ότι ανάλυση των πραγματικών περιστατικών, των στοιχείων που επηρεάζουν ε, στην πραγματικότητα την παρουσία των κοριτσιών στο σχολείο ή το ζήτημα της παρουσίας των διδασκόντων, ε, είναι ένα σοβαρό ζήτημα και πρέπει να εξεταστεί μόνο κατά περίπτωση και κατά κράτο. Ε, η Επιτροπή κατά την άποψή μου τώρα να λάβει μια πολύ σημαντική ε, δουλειά που είναι η επαλήθευση των μεθοδολογικών κύκλων για το Project Cycle Management όπου ενσωματώνει ένα μεθοδολογικό κύκλο για τους κύκλους πώς αξιολογούνται οι δείκτες, πώς χρησιμοποιούνται. Και είναι δείκτες όχι δικοί μας, είναι δείκτες πορείς στο ίδιο το κράτος και πώς μπορούμε ε, σε έναν τομεακό διάλογο με τη χώρα να τοποθετηθούμε ε, ως προς την αξία των δικτών. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ε, δουλειά για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το οπλοστάσιο που έχουν τα κράτη και να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν καλύτερα τους δείκτες. Επίσης αναφερθήκατε στους, ε, σε, σε πρόσθετα στοιχεία αριθμητικά. Υπάρχουν στα στοιχεία που έχει καταγράψει ανακράτος στο ελεγκτικό συνέδριο. Αντίρρηση από πλευρά μας δεν υπάρχει. Μπορούμε να σας τα διαθέσουμε τα αριθμητικά αυτά στοιχεία. Ε, υπάρχουν ενδεχομένω πιο πολλά στοιχεία στις εκθέσεις χώρα που δεν έχουν ασωματωθεί στη συνολική έκθεση. Επίσης το εξειδικευμένο προσωπικό Βλέπω ότι σας απασχολεί. Πιστεύω ότι τώρα που η Επιτροπή έχει, θα έλεγα, μια συνολική έποψη για το προσωπικό που αναλαμβάνει δράση από την προηγούμενη χρονιά από 1η Δεκεμβρίου και λειτουργική εικόνα της λειτουργικής ε, παρουσίας των αντιπροσωπιών μας μπορούμε, και αυτή είναι και η πρόθεσή μας, να επαναπροσδιορίσουμε, να εξισορροπήσουμε το προσωπικό μας στις αντιπροσωπείες ε, κατά τρόπον ώστε να, αλλάξουν, ε, να, λήξουν, να αλλάξουν οι ισορροπίες ως προς τη βοήθεια που προσφέρεται στα κράτη, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και ως προς την, ε, τις δεξιότητες που θα έχει το προσωπικό στην κάθε αντιπροσωπεία. Δηλαδή το άτομο που έχει τις κατάλληλες δεξιότητες το κατάλληλο κράτος. Ε, ασφαλώς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας για το θέμα αυτό. Είναι πολύ μεγάλη σημασία και για μας όπως και για σας και με πολύ μεγάλη χαρά προσμένω τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση. Ο κύριος Οντί έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να χαιρετήσω την ποιότητα της έκθεσης, της πληροφορίες που περιλαμβάνει για τη δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων, των δημόσιων αυτών κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. θα ήθελα να κάνω μια πρόταση, ίσως σας φανεί κάπως Ερετική αυτή τη στιγμή. Διερωτώ με λοιπόν, εάν υπάρχει αν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να γίνει μια συνολική επαλήθευση για ορισμένου τομεί των δημοσίων δαπανών ω προ την παρουσία ε, των τριών ε, επιπέδων εξουσίας για τις ε, αμυντικές δαπάνες, την πολιτική διπλωματία και ούτω καθεξής, εξωτερική πολιτική διπλωματία και ούτω καθεξής. Αυτά για το τρία επίπεδα, δηλαδή ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό. Και αυτό βλέπουμε και σαν ε, τρόπο αξιολόγησης χρηματοδότησης ανάπτυξης στα 113 δισεκατομμύρια, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, τα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης. Φαίνεται δηλαδή να έχουμε πληθώρα παρεμβάσεων που πολλαπλασιάζονται διαρκώς και διερωτώ εάν σε συνεργασία και με τα κράτη-μέλη υπάρχει δυνατότητα να αναπτύξουμε μία, ε, έναν έλεγχο για το θέμα της ανάπτυξης έτσι ώστε να έχουμε υπόψη ποια παρέμβαση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έλεγα όχι όμως ποσοτικά δηλαδή από πλευράς της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράγοντα, έτσι ώστε να έχουμε μια συνολική θεώρηση. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω καλά είναι υπάρχει κάποια αξία που προσθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την παρέμβαση. Πέραν αυτών των παρεμβάσεων υπάρχει η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Και αυτό λέω γιατί έχω αναλάβει ως συγκεκριτή αναθεώρηση του, της λειτουργίας του ε, τρέχοντος 7ου προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα. Διερωτώμαστε όμως αν τελικά αυτά τα προγράμματα προσφέρουν κάτι επιπλέον. Ευχαριστώ κυρία Κρίσλα. Ευχαριστώ. Και εγώ καλωσορίζω την έκθεση, είναι πολύ σημαντική, πολύ ενδιαφέρουσα ε, περιέχει στοιχεία τα οποία δεν είχαμε ε, λάβει μέχρι τώρα. Ο κόσμος αλλάζει αργά, ελπίζουμε ότι πηγαίνει προς την καλή κατεύθυνση και θα ήθελα συγκεκριμένα για την εκπαίδευση να ρωτήσω εάν έχουμε συγκεκριμένη εικόνα του πόσους δασκάλους χρηματοδοτούμε. Πώς, με ποιο τρόπο υπάρχουν αριθμοί λογαριασμού, ο οποίος καταθέτουμε τα χρήματα, πώς γίνεται. Γιατί βέβαια θα ήθελα ο δάσκαλο στην κάθε χώρα να είναι αυτό ο οποίο εισπράττει τα λεφτά και όχι κάποιο σύμβουλος ή ενδιάμεσο παράγοντα. Αυτή η δημοσιονομική βοήθεια στο δάσκαλο πρέπει να πηγαίνει. Ε, μην ξεχνάμε ότι αυτή η δημοσιονομική ενίσχυση ε, έχει κάπως εχει καπω δυσφημιστει ε, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν και θέλω να πω δεν έχουμε και πολλέ εναλλακτικέ. Μας περιπτώσει με ενδιαφέρει άμεσα να καταβάλλονται τα κονδύλια και να έχουμε και τη σχετική ενημέρωση. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Αγιάλα Σέντερ. Sí, gracias, presidente, Sí, en la misma línea que que mi compañera señora Gresle, eh, ayer. Εχθές μιλούσαμε για το θέμα της ενίσχυσης του προϋπολογισμού Εγώ δεν συμφωνούσα με αυτήν τη σύγκριση που έκανε μεταξύ κρατών μελών και τρίτων ε, χωρών για τα θέματα ανάπτυξης και ρωτώ την Κομισιόν ήρθαμε πλέον εδώ στο θέμα της δημοσιονομικής ενίσχυσης και το θέμα της εκπαίδευσης ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά αυτό το τελικό τελικά αυτό το θετικό στοιχείο στο οποίο καταλήξαμε ότι η δημοσιονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί σωστά και όσον αφορά δηλαδή στον έλεγχο μετά κλπ. Παρόλα αυτά όμως πέρα από τη λογιστική δαπάνη, αν δηλαδή ξοδεύεται σωστά από λογιστικής πλευράς το χρήμα, θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το άλλο αποτέλεσμα που δεν είναι το λογιστικό. Και κυρίως για την Βόρειο Αφρική το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Όλι Ρεν. Αν υπήρχαν λοιπόν δυσλειτουργίες που οδηγούσαν τον κόσμο να ξεσηκώνεται, τους λαούς να ξεσηκώνονται με το δίκιο τους. Ρωτώ την Κομισιόν, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση σε αυτό που μας προτείνει το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και στο δικό μας προβληματισμό για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και αν προβλέπουμε κάποια δυνατότητα. Για την εκπαίδευση τώρα υπάρχουν δύο στοιχεία που τα θεωρώ σημαντικά. Ρωτώ. Το λέει το λεκτικό συνέδριο. Δεν ξέρω αν έχουν παραπάνω πληροφορίες στο ρωτώ και στην Κομισιόν. Οι δείκτες για την εκπαίδευση δεν φαίνεται να επαρκούν είναι περισσότερο, χάνονται μέσα στις, ε, στους δείκτες για τη γενική εργασία. Τώρα για τις εξωτερικές υπηρεσίες της Ένωσης, για το μέλλον τουλάχιστον, ότι δεν είναι εξοπλισμένες ε, σε ανθρώπινους ε, πόρους αλλά και εντολή για τα θέματα εκπαίδευσης. και όσον αφορά στην αναπτυξιακή βοήθεια πώς σκέφτεται η Κομισιόν να ενισχύσει αυτές τις αντιπροσωπείες ώστε να είναι έτοιμες για το διάλογο αλλά και για την άσκηση πολιτικής σε εκπαιδευτικά θέματα με αυτά αποτελέσματα. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Euh, euh, Θέλω να επανέλθω λίγο σε αυτό που είπα στην αρχή της παρέμβασής μου της πρώτης και να σχολιάσω και κάποια από τα θέματα που ετέθησαν. Νομίζω ότι πηγαίνουμε πολύ καλά ε, και συμφωνούμε και ο Επιτροπός Πίμπαλξ το είπε και μάλιστα και στις δύο πράσινες ε, βίβλους και για την ανάπτυξη και για τη δημοσιονομική βοήθεια θέλει να είναι προσανατολισμένη στις προσπάθειες και στα αποτελέσματα φυσικά, αλλά θέλει να σκεφτούμε και σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν προγραμματίζουμε τη βοήθειά μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί οι ροές χρημάτων προς τις χώρες αυτές, θα έλεγα η ροή βοήθειας είναι ένα πυροελάχιστο πραγματικά τμήμα όλων των ροών χρημάτων που επενδύονται σε καθεμία από τις χώρες. Από το, ε, πάμε, είναι το ένα σε μια κλίμακα των 20 θα έλεγα. Επομένως, εντάξει, ε, το έχουμε θέσει και εμείς το ερώτημα και μπορούμε να το σκεφτούμε πώς μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε τη βοήθεια αυτή για να επηρεάσουμε σε σχέση με τα πραγματικά προβλήματα. Εμείς νομίζουμε ότι η δημοσιονομική στήριξη, το είπε πολύ καλά και το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί δεν θέτει υποαμφισβήτηση αμφισβήτηση ε, την στήριξη μέσω του προπολογισμού. Αυτό το οποίο σωστά αμφισβητεί είναι ε, πώς, ή μάλλον ε, μας θέτει το εξής ερώτημα, πώς Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τα κατάλληλα ποσά, τα επαρκή ποσά για την επίτευξη των στόχων και κυρίω ποιοι είναι οι δείκτε που θα χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε ότι πράγματι υπάρχουν αποτελέσματα σε τομεακό επίπεδο. Πανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν. Δεν είμαστε οι κύριοι του έργου εμείς, ε, είμαστε, ε, μάλλον οι χώρες είναι αυτές. Εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε με τη δημοσιονομική μας βοήθεια και ίσως θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε ακριβώς με το διάλογο για τις πολιτικές και για τους δείκτες. Η χώρα όμως θα ορίσει τους δείκτες αυτούς και τους στόχους της πολιτικής της, το όραμα που έχει κάθε χώρα για την επόμενη πενταετία, δεκαπενταετία, εικοσαετία. Αν λοιπόν έχουμε έναν σωστό διάλογο σε επίπεδο κυβέρνηση και όχι μόνο σε επίπεδο κυβέρνηση, είναι σημαντικό όλοι οι φορείς να συμμετάσχουν στην προσπάθεια τα εθνικά κοινοβούλια, κοινωνία των πολιτών κτλ. Είναι πολύ σημαντικό και εμείς προς τα εκεί παροτρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να ιδιοποιηθούν συνολικά οι χώρες και να έχουν και τους κατάλληλους δείκτες για αυτήν την προσπάθεια. Εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και έχουμε ξεκινήσει ε, να το κάνουμε, αλλά καταλάβαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο δραστήριοι. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι διαθέτουμε εργαλεία για τις αντιπροσωπείες ώστε να μπορούν με αποτελεσματικό τρόπο να πραγματοποιήσουν το διάλογο αυτό για τις πολιτικές και να κατανοήσουν ακριβώς γιατί αποτελέσματα μιλάμε. Μιλάμε για βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Τις προάλλες κάποιος μου μιλούσε για την δικτατορία του βραχυπρόθεσμου αποτέλεσματος και αυτό πραγματικά πρέπει να το προσέξουμε. Όλοι θέλουμε να δούμε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, να δούμε γρήγορα αποτελέσματα. Προσοχή όμως αυτά δεν θα πρέπει να εμποδίσουν ε, το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, γιατί η ανάπτυξη είναι μακρόπνοη προσπάθεια και πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνέπεια και συνεκτικότητα. Πώς ε, καταβάλουμε τους μισθούς, τους εκπαιδευτικούς. Πράγματι, πολύ ευστόχο και σωστό το ερώτημα. Γιατί συχνά έχει ως αποτέλεσμα τις συχνές απουσίες των εκπαιδευτικών. Δεν είμαι εμπειρογνώμος στον τομέα αυτό, αλλά έχω ακούσει Κάποιος να λένε ότι μέσω του κινητού, της κινητής τηλεφωνίας, μπορούσαν να καταθέτουν τους μισθούς ε, στους ε, εκπαιδευτικούς αυτού. Και δεν ζητούσαν τίποτε άλλο. Υπάρχουν κάποιες καινοτόμες λύσεις που τις θαυμάζω θα έλεγα. Και εγώ είμαι ακόμα στην εποχή της γραφής Όλα αυτά που γίνονται πραγματικά μου φαίνονται σχεδόν σαν θαύμα. Αλλά ε, αυτή τη στιγμή ε, με κάποιες χώρες μελετούμε αυτού του είδους τις καινοτομίες που πραγματικά είναι ιδιαίτερα ε, ελπιδοφόρες και υπόσχονται πολλά για την καταπολέμηση του απουσιασμού, των συχνών απουσιών. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιες ερωτήσεις. Α, ναι για τους συναδέλφους που είναι σε αντιπροσωπείε ε, και τις δυνατότητε ε, ε, Η τις ικανότητε μου πραγματικά έχει τονίσει το ζήτημα τη ποιότητα των επιχειρησεων αντευκο η διευθυνση μου πραγματικα εχει τονισει το ζητημα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, ότι πρέπει ίσως οι συμπεριγνώμενες όχι να είναι την αντιπροσωπεία, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Στη Ζιμπάμπουε, στην αντιπροσωπεία, είχα ένα περιφερειακό εμπειρογνώμονα για τη θέματα τη υγεία στη Ζιμπάμπουε, ο οποίο κάλυπτε όλη την περιοχή. Και αυτή είναι μια δυνατότητα την οποία μπορούμε να ε, αξιοποιήσουμε ενδεχομένω, αν δεν έχουμε παρκή προσωπικό σε κάθε χώρα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ε, την κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων από την περιφέρεια, από την περιοχή. Είναι θέματα όλα αυτά τα οποία είναι υπό εξέταση μαζί με το γενικό ε, διευθυντή μας και τον άλλο επίτροπο τα συζητούμε και είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Ευχαριστώ. Το ελεκτικό συνέδριο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, δύο από τα ερωτήματα αφορούσαν το ελεκτικό συνέδριο και θα ξεκινήσω με αυτό του κυρίου Οντί. Πάντοτε υπάρχει ένα σκεπτικισμό, μια επιφυλακτικότητα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε μια, ένα μεγάλο κοινό ε, έλεγχο ε, με όλους τους 27 φορείς. Τώρα, ε, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους εθνικούς ελεγκτικούς φορείς ε, και στον τομέα της ανάπτυξης. Έχουμε ένα πλαίσιο, ΧΟΑΠ λέγεται. Εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο συμμετέχουμε ενεργά και υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία ενεργά παρέχουν αναπτυξιακή βοήθεια ε, σε ανεψόμενες χώρες ε, που συμμετέχουν επίσης ενεργά, όχι μόνο 27 χώρες μέλη. Και βέβαια δεν είναι μυστικό να πούμε ότι κάποια πράγματα τα οποία επικρίνουμε ε, στην Κομισιόν τα επικρίνουμε ίσως και από τους εθνικούς, τους εθνικούς φορείς και στις κυβερνήσεις. Το βλέπετε νομίζω πολλές φορές ε, στις ε, εκθέσεις μας. Υπάρχουν κάποιες φορές και ρητές ε, απευθείας αναφορές. Και κάποτε υπάρχουν τα ίδια συμπεράσματα τα οποία συνάγουν. Εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο είμαστε εδώ για να δίνουμε συμβουλές στην Κομισιόν. σε ό,τι αφορά ιδίως τις ε, εκθέσεις ελέγχου στον τομέα των επιδόσεων, της απόδοσης. Δεν υπάρχει βέβαια μία συνταγή για όλους, η ίδια για όλους. Αν θα είναι η γενική δημοσιονομική υποστήριξη, η τομεακή ή η βοήθεια μέσω έργων. Δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι το καλύτερο. Ε, κάθε φορά ε, πρέπει να εξατομικεύσουμε ανάλογα με τη χώρα εν μέρη είμαστε, ε, μάλλον εν γέννη είμαστε υπέρ της δημοσιονομικής στήριξη, της βοήθειας μέσω του προϋπολογισμού που είναι και ένας τρόπος για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση στη χώρα και να υπάρχει ε, ιδιοποίηση της προσπάθειας από την ίδια τη χώρα. Συμφωνώ και με τη δημιουργία υποδομών και τη δημιουργία ικανοτήτων για την οποία μίλησε η Κομισιό. Πάντοτε όμως είναι θέμα χώρας. Υπάρχουν χώρε που δεν είναι όριμε θα έλεγα, για μια τέτοια βοήθεια. Σε ό,τι αφορά τους δείκτε, αν κατάλαβα καλά, ε, με ρωτήσατε αν οι δείκτε είναι επαρκεί και αξιόπιστοι. Κυρία Γιάλα, νομίζω, με ρώτησε. Κοιτάξτε, κατά πόσον είναι επαρκεί οι δείκτε. Στην έκθεση εκφράσαμε κάποια ε, κριτική για τους δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης. Νομίζουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητε για να μετρήσουμε την ποιότητα. Δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί η ποιότητα γενικά. Πάντως ε, υπάρχουν ε, κάποιες ε, ιδέες, όχι και τόσο λαμπρές, αλλά αν υπάρχουν καλές ιδέες είναι και πολύ δαπανηρές. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα, φαίνεται η Κομισιόν να μην εκμεταλλεύτηκε όλες τις δυνατότητες για τη μέτρηση της ποιότητας. Ενίοτε και μάλιστα επισκέφθηκα μια αντιπροσωπεία, μια αποστολή στο Νεπάλ στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου και πραγματικά ξεπλάγει. Δεν ήταν τόσο ε, σφάλμα της Επιτροπής αλλά από τους άλλους δωρητές. Οι δείκτες για τις διάφορες δόσεις της βοήθειας ήταν προσανατολισμένη πιο πολύ στις διαδικασίες και όχι στην, στο αποτέλεσμα, το απτό. Θα πρέπει να το δούμε το θέμα της επάρκειας. Και έχουμε και μία συζήτηση διαρκή με την Κομισιόν για τη δομή των δικτών στη γενική υποστήριξη μέσω προπολογισμού. Παράγραφος 83 γάμα συγκεκριμένα. Είναι πρόκληση. Είναι θέμα ακόμη για την Κομισιόν. Και στη συζήτηση για την πράσινη βίβλο πρέπει να δούμε και τα τομεακά ζητήματα. Νομίζουμε ότι πρέπει να καλυφθούν καλύτερα ή καλύπτονται καλύτερα μέσω της γενικής δημοσιονομικής στήριξης αν λάβετε υπόψη τη σημασία που έχει η εκπαίδευση, το να υπάρχουν τρει-τέσσερι μόνο δείκτε για τη βελτίωση τη εκπαίδευση στου δείκτε για τη γενική δημοσιονομική στήριξη δεν είναι επαρκέ. Σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των δικτών, και αυτό είναι ένα μείζον θέμα, στην έκθεση έχουμε επαναλάβει και εμεί ότι ε, Ω ελεγκτικό συνέδριο χρειαστήκε να βασιστούμε πολλές φορές στα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας και κατά την άποψή μας είπαμε ότι παρά τη στήριξη των δωρητών τα εθνικά στατιστικά στοιχεία των χωρών ε, δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε αξιόπιστα. Υπάρχουν και κάποια παραδείγματα, παραδείγματο χάρη διαφορέ μεταξύ των εθνικών στατιστικών για τους σκοπούς εκπαίδευσης και της έρευνας για την οικοκυριά. Μεγάλες, τεράστιε διαφορές στις δύο αυτές περιπτώσεις για τον αριθμό των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο. Πάλι από τη χώρα που επισκέφθηκα το Νεπάλ, ή το γνωρίζετε αυτό. για την εγγραφή στο σχολείο, κατά πόσον πηγαίνουν ή όχι στο σχολείο τα παιδιά. Την πρώτη μέρα ε, γράφονται, ε, αλλά από εκεί και πέρα κανεί δεν ενδιαφέρει να παρακολουθούν τα μαθήματα. Άρα μένει. Το πρόβλημα ισχύει ακόμα. Σίγουρα δεν είναι η Κομισιόν ε, αυτή η οποία θα πρέπει να αναλάβει και να θέσει σε πέρας όλα τα θέματα της βελτίωσης. Η κυρία Γιάλα. Σε σχέση με αυτό που μας είπε η Διευθύντρια για την ποιότητα του προσωπικού στις αντιπροσωπείες, ευχαριστώ που έχει κατά νου την βελτίωση των ικανοτήτων διότι το προφίλ των υπαλλήλων που καταλήγει στις ε, αντιπροσωπείες ε, δεν είναι πάντα ένα προφίλ ε, εξειδικευμένο στην παιδεία είναι συνήθως νομικοί, έχουν άλλες ειδικότητες, ο, ο χώρος της παιδείας είναι εντελώς διαφορετικός, είναι θεμελιώδες λοιπόν, είναι βασικό <coughs> το να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και εμπειρογνώμονες σε θέματα παιδείας. διότι στα 4-5 χρόνια που κρατάει μια θητεία δεν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας σε αυτόν τον τομέα. Ο συνάδελφος Τάις ε, για να ολοκληρώνει ευχαριστώ πρόεδρε τελειώνω δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή, ήταν πολύ καλή όλη αυτή η συζήτηση όπως και η απάντηση της Κομισιόν και ευχαριστώ και για την συμπλήρωση των ε, πληροφοριών εκ μέρους του ελεγκτικού συνεδρίου θα εξετάσουμε χώρα με χώρα. Η κυρία Γκρέσλε το είπε σαφέστατα και στην τοποθέτηση της. Η δημοσιονομική βοήθεια είναι μία μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιήσαμε. Το μόνο πρόβλημα είναι να πάει αυτή η βοήθεια εκεί που πρέπει να πάει και να χρησιμοποιηθεί σωστά. Η Κομισιόν είχε την ε, καλοσύνη και την ευχαριστώ για την πράσινη βίβλο και εμείς οι ευρωβουλευτές πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας διότι ο κύριος ε, Κέρενς συζητά αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, την δημοσιονομική βοήθεια. Και βέβαια τα επιχειρήματα που μας διαβιβάζει το ελεκτικό συνέδριο είναι εξαιρετικά. δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις για αυτό το σημείο, πάω στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της Όλα. Την παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων και τις δραστηριότητε για το 2009. Δίνω το λόγο στα δύο στελέχη της Επιτροπής Εποπτείας για να παρουσιάσουν την έκθεση. Είναι παρόντες εδώ η κυρία Ράιτ και ο Λουίς Λόπες Σάντς Αράγχουες. Ποιος από τους δύο θέλει το λόγο? Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω Εκ μέρους της Πρόεδρου, κυρία Στέατο και της Συμβουλευτικής Επιτροπής, και τις γραμματείας μας. Θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Επιτροπής σας που προσέφεραν στον κύριο Σανζαλάν Λουας Λόκπες και την υποφανομένη την ευκαιρία να συστήσουμε τα θέματα αυτά και να σας παρουσιάσουμε την ε, έκθεσή μας και τις δραστηριότητες από τον Ιούνιο 2009 στο Δεκέμβριο του 2010. Ήταν μια πολύ επικοδομητική περίοδος, δημιουργική περίοδος για την Επιτροπή μας. Ασχολήθηκε μια σειρά από ζητήματα ε, συντάξαμε πέντε γνωμοδοτήσεις και ασχοληθήκαμε και με την, διαδικασία της, ε, του διορισμού νέου Γενικού Διευθυντή της Όλαφ. Καλωσορίζουμε το διορισμό του κύριου Τζοβάνι Κέσλερ για τη διάρκεια της δικής μας ε, θητείας ε, στη θέση αυτή και έχουμε αρχίσει ήδη τη συνεργασία μαζί τους σε επικοδομητικούς όρους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, λοιπόν, ε, η Επιτροπή μας υλοποίησε τον κύριο στόχο της, που ήταν η παρακολούθηση της ε, υλοποίησης του ερευνητικού έργου της ΟΛΑΦ και της ολοκλήρωση των ε, ανακρίσεων. Η Επιτροπή Αποπτίας ιδιαίτερη προσοχή έδωσε στην παρακολούθηση από πλευράς της Όλαφ και την συνέχεια που έδινε η Όλαφ στις δικές μας συστάσεις, κυρίως ως προς τη διάρκεια των ανακρίσεων και την απουσία σαφών λόγων για κάποια ενδεχόμενη καθυστέρηση. Παρακολουθήσα μια σειρά από ανακρίσεις, 164 συγκεκριμένα, για να καταθέσουμε συγκεκριμένες ε, και καινοτόμες προτάσεις προς την Όλαφ, προκειμένου να τη στηρίξουμε στην προσπάθεια για αλλαγή του συστήματος ανακρίσεων και ταυτόχρονα ε, ιδιαίτερα μας ενδιέφερε να δούμε από πλευρά της Όλαφ μια αποφασιστική δράση σε ορισμένες και περίπλοκες περιπτώσεις, ε, στόχους και προτεραιότητες στη δουλειά της και επαγγελματική ε, λειτουργία στηριζόμενη σε κάποιο εγχειρίδιο. Δυστυχώς όμως, έχουμε απογοητευτεί προς αυτό, δεν ακολούθησε τις συστάσεις μας η Όλαφ. Επίσης, στο τέλος, ε, το τελευταίο αυτό τμήμα της εντολής μας, με επιμονή τοποθετηθήκαμε στο θέμα αυτό και το υπογραμμίσαμε, υπογράψαμε τη σημασία του για τον ακριτικό έργο της Όλαφ και την ανεξαρτησία της. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ο χρόνο αφιερώσαμε, το μέγιστο χρόνο αφιερώσαμε ως προς την εφαρμογή του κανονισμού 1073 του 99 που αφορά την ΟΛΑΒ, Θεωρούμε ότι το έγγραφο μελέτης του Επιτρόπου Σεμέτα που ε, ορίζει τις συστάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ σημαντικό, το παρακολουθήσαμε, το μελετήσαμε, εμπλακήκαμε στη συζήτηση και όχι μόνο. θεωρούμε ότι εμπλέκονται και τα κρατη θα πρέπει μάλλον να εμπλέκονται και τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται από αυτό. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διαφυλαχθούν οι εξουσίε ανακριτικέ τη Όλαφ, να, να ενισχυθούν όπου είναι δυνατόν και να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία τη. Θα δείτε τα απόγευμα παρουσίαση από τον Επίτροπο Σεμέτα του νέου κειμένου για τη μεταρρύθμιση του λόγου κανονισμού που δεν είχαμε εμεί ακόμη την ευκαιρία να δούμε και όσο μπορούμε να σχολιάσουμε. Πλην όμω η Επιτροπή μα μπορεί, πιστεύω, ε, να συνοψίσει το έργο της ως εξής. Καλώς ορίζουμε μεγάλο κομμάτι αυτών των προτάσεων και των μηχανισμών που προτάσσονται για τη λειτουργία του μηχανισμού ροής πληροφοριών προς την Επιτροπή μας κατά τη διάρκεια μιας ανακριτικής διαδικασίας που θα επιτρέπει στην Επιτροπή μας να εξασφαλίζει την, ε, να διασφαλίζει μάλλον την ανεξαρτησία αυτής της ανακριτικής δράσης και λειτουργίας. Η Επιτροπή μας ωστόσο εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν ε, λήφθησαν υπόψη οι συστάσεις μας για τη μεταρρύθμιση και για τις προτάσεις ε, τις σχετικές με τις ιστορικές και εξωτερικές ε, ανακρίσεις και έρευνες και ιδιαίτερα θεωρούμε ότι η προτεραιότητα, ε, ο προσδεσμός προτεραιότητων αναϋπόθεση θα πρέπει να ενσωματωθεί και βέβαια ο κανόνας de minimis εισάγεται μέσα στο νέο κανονισμό. Η συνθήκη της Λισαβόνας τώρα επιτρέπει μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων και εθνικών δικαστικών αρχών. Η Επιτροπή ιδιαίτερως υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ισχύουσα αρχιτεκτονική δομή αυτού του συστήματος θα πρέπει να διαφυλαχθεί, η ανεξαρτησία δηλαδή τη Όλεφ μέσα στην Επιτροπή, ανεξαρτησία του Γενικού Διευθυντή και τη ανακριτική λειτουργία. παρακολούθηση από τη δική μα Επιτροπή τη ανεξαρτησία τη Όλαφ ε, και από εξωτερικού οργανισμού. Ε, είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διαφυλαχθούν στο σύνολό τους. Από την άλλη, ωστόσο, η Επιτροπή μας εκφράζει την ανησυχία της για την ε, πρόταση ε, περί θέσπισης ενός συμβούλου επιτήρησης που θα ενισχύσει το γραφειοκρατικό φόρτο και θα προξενήσει καθυστερήσεις στην παραγωγή του έργου. Και η παρακολούθηση από μια επιτροπή της ε, του έργου και των υποθέσεων που ερευνάει όλα πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε βραδιπορίε και ενδεχομένω να επηρεάσει και την ανεξαρτησία τη ε, ανακριτική λειτουργία τη Όλαφ. Η Επιτροπή μα βέβαια θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στις, ε, στους φακέλους και τις υποθέσεις που έχει μελετήσει η Όλαφ για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε ε, ότι όντως και η αποτελεσματικότητα και η αποτελεσματικότητα αλλά και η ανεξαρτησία στην ε, λειτουργία της Όλαφ έχουν διαφυλαχθεί. Επίσης ε, προειδοποιούμε για τον ενδεχόμενο κείμενο υπερβολικών ρυθμιστικών, ρυθμίσ, ε, κανονιστικών ρυθμίσεων εις βάρος του έργου της Όλαφ και θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα στο μέλλον, εάν εισαχθούν τέτοιοι όροι, να ε, εξασφαλιστεί και δυνατότητα για εισαγωγή ενδίκων μέσων σε αποφάσεις της Όλαφ. Ε, πάντως θέλουμε να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, η ηγεσία της Όλαφ θεωρούμε ότι θα πρέπει να καθοδηγεί τις ε, ανακρίσεις και την ταχύτατη διεξαγωγή, την τάχιστη δυνατή διεξαγωγή και ολοκλήρωση αυτών. Επίσης θεωρούμε ότι ο νέος Γενικός Διευθυντής της Όλαφ θα πρέπει να έχει επαρκή χρόνο στη διάθεσή του ώστε να ε, να διαβουλεύεται για τα θέματα αυτά, να δίνει τη γνώμη του. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση που ε, είχαμε εμεί τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε, είχε μέσα σε 10 μέρε τη δυνατότητα να καταθέσει 11 διαφορετικέ νομοδοτήσει. Η Επιτροπή μα παρακολουθεί λοιπόν τη διαδικασία τη αναθεώρηση και θα περιμένω να ακούσω σήμερα τον Επίτροπο Σεμέτα και τι προτάσει του. Επίσης εξετάσαμε και το θέμα του προγραμματισμού ε, στις έρευνες. Εξετάσαμε δειγματοληπτικά 40 υποθέσεις ε, από τις διευθύνσεις Α και Β για να δούμε κατά πόσο και σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός βοηθά την Όλαφ για να διεξαγάγει τις έρευνές της όπως ε, αναφέρεται και στην έκθεση πεπραγμένων για το 2008-2009 η εξέταση του σχεδιασμού και η στρατηγική κατεύθυνση των υποθέσεων είναι ένα απόσπαστο τμήμα του έργου μας για την παρακολούθηση των ερευνών ώστε ε, να διασφαλίσουμε ότι η Όλαφ ε, εργάζεται αποτελεσματικά και αξιοποιεί ε, με τον καλύτερο τρόπο του περιορισμένου πόρους τη. Και κατέληξαμε στο συμπέρασμα ότι μπορεί ο σχεδιασμός να βελτιωθεί σημαντικά σε όλους του επιχειρησιακούς τομείς για τρεις βασικούς στόχου. Πρώτον, για να επικεντρωθούν όλοι οι ερευνητέ, ο τη μονάδα και οι υπόλοιποι στην στο στόχο. Έπειτα να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα για την έρευνα, να αποδοθούν επίσης οι κατάλληλοι πόροι για την έρευνα και τρίτον για να υπάρχει και ένα πλαίσιο βάσει το οποίο θα μπορούν να εξετάζουν οι διευθυντές πώς προχωρά η έρευνα, αν υπήρξαν ε, αχρίαστες καθυστερήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ή αν άλλαξε η κατεύθυνση έρευνα σε σχέση με την αρχική εκτίμηση και αν θα πρέπει να διακοπεί όχι έρευνα. Η Επιτροπή συνιστά να υπάρχει ένα πρότυπο, ε, ένα υπόδειγμα από την Όλαφ για οποιοδήποτε σχέδιο έρευνας. Σίγουρα ποτέ δεν είναι ταυτόσιμες δύο έρευνες, αλλά κάποιες φορές ε, ή μάλλον σε όλα τα σχέδια πρέπει να υπάρχουν κάποιες κοινέ πτυχές, ε, κάποια κοινά σημεία. Και βέβαια αυτά θα διαφέρουν στη φάση της αξιολόγησης από την φάση της έναρξης της έρευνας. Και θεωρούμε ότι κάθε σχέδιο θα πρέπει να το εξετάζει να εξετάζεται αφού θα έχει ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο για έναρξη μιας ε, έρευνας. Είναι ένα δυναμικό έγγραφο, ξέρουμε, ε, το σχέδιο αυτό. Επίσης, θα πρέπει από το σχέδιο να μπορεί και ο ερευνητή και ο επικεφαλής μονάδας και ο διευθυντής να βλέπει κατά πόσον η έρευνα προχωρεί ομαλά, υπάρχουν δυσκολίες. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το σχέδιο να μπορεί ο επικεφαλής ομάδα να δει σε ποια φάση έχει φτάσει η έρευνα, αν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, αν θα πρέπει να αλλάξουν τα χρονοδιαγράμματα, αν υπάρξουν νέε προτεραιότητε, αν έχουν εκτελεστεί τα καθήκοντα από κάθε ερευνητή ή κατά πόσον έχουν ε, οι ερευνητέ προγραμματισμένα καθήκοντα για τι επόμενε εβδομάδε. Και πριν την λήξη τη εντολή, η Επιτροπή θα δει κατά πόσον και σε ποιο βαθμό έχουν εφαρμοστεί από τον Όλαφ οι συστάσει ε, για το σχεδιασμό των ερευνών. Μία άλλη σημαντική γνωμοδότηση που δημοσίευσε η Επιτροπή σε αυτή την περίοδο αφορούσε τις ε, εγγυήσει, ε, μάλλον το σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις διαδικαστικές εγγυήσει. Ο κύριος Λόπεθ θα σας πει τα σχετικά. Πέραν αυτού του έργου, εξετάσαμε το σχέδιο προπολογισμού τη Όλαφ για την περίοδο 2010-2011, Κάναμε την τακτική παρακολούθηση των νέων υποθέσεων και εξετάσαμε και τι τελικέ εκθέσει για τι διάφορε υποθέσει και τι συστάσει που έχει υποβάλει η μονάδα ΓΑΜΑ 1 σε εθνικέ δικαστικέ αρχέ για τις ε, υποθέσει των οποίων έχει επιληφθεί για περαιτέρω δράση. Τα συμπεράσματά μα σε σχέση με την τελευταία περίπτωση ήταν ότι αυτέ οι εκθέσει θα μπορούσαν να είναι πιο συνεκτικέ και σαφέστερες και αυτό που θέλουμε και προτιθέμεθα να κάνουμε στου επόμενου μήνε είναι να εξετάσουμε την έκβαση αυτών των διαβάσεων για να δούμε κατά πόσον θα μπορούσε η Όλαφ να κάνει και κάτι ακόμα ώστε να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα όπου αυτό είναι δυνατόν. Πανέρχομαι στον προπολογισμό τη Όλαφ. Ακούσαμε με χαρά ε, τη δήλωση του κυρίου Κέσλε στην Επιτροπή Έλεγχου του Προπολογισμού κατά τη διαδικασία επιλογή ε, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή ότι θα ήθελε το 5% του προσωπικού τη Όλαφ να εργάζεται στι έρευνε. Ελπίζουμε να τηρήσει την δέσμευσή του. Φυσικά συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε, μάλλον εργαζόμαστε εντατικά στην παρακολούθηση των υποθέσεων. Ε, θέλουμε μια μερόληπτη Όλαφ και θέλουμε να το διασφαλίσουμε αυτό και κοιτούμε τώρα ε, τις εννιάμινες εκθέσεις αλλά και κάποιες υποθέσεις ε, ε, που έχουν περάσει τα τέσσερα χρόνια διάρκειας και κατ' αίτημα της ίδιας της Όλαφ εξετάζουμε την πρόσβαση της Όλαφ σε δεδομένα του προσωπικού, του εσωτερικού προσωπικού, τα οποία διατηρεί η Κομισιόν και τα οποία μπορεί να σχετίζονται με τις εσωτερικές έρευνες. Θα συνεχίσουμε όμως να εργαζόμαστε και για την μεταρρύθμιση του κανονισμού 1073. Κατά το τελευταίο έτος εντολής μας θα εξετάσουμε το έργο που έχει γίνει στη διάρκεια της εξαετίας και θα δούμε κατά πόσον η Όλαφ έχει ακολουθήσει τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις γνωμοδοτήσεις μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Ράι, το άλλος εκπρόσωπος, ο κύριος Λόπες Σάντσαράνκουες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως το ανέφερε και η κυρία Ράιτ, ε, θα αναφερθώ στο 5210 της Επιτροπής Εποπτείας, η οποία βρίσκεται ως παράρτημα στην έκθεση δραστηριοτήτων. Και θα αναφερθώ στους λόγους που οδήγησαν την Επιτροπή να επεξεργαστεί αυτή τη γνωμοδότηση, τη μεθοδολογία, τους στόχους και τις συγκεκριμένες προτάσεις αυτής της γνωμοδότησης για τους λόγους. Πρώτο, κάθε έκθεση, ερευνητική έκθεση που μπορεί να πάει σε κυρώσεις διοικητικές, ε, πειθαρχικές ή ποινικές, ε, πρέπει να είναι μία διαδικασία που να σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης, μία διαδικασία που να πληρεί όλες τις εγγύησεις, διότι αυτό οδηγεί και στην τελική αποτελεσματικότητα των ερευνών και έχει επιπτώσεις στους οργανισμούς που ασκούν την έρευνα, στην αξιοπιστία τους και επίσης ε, διασφαλίζει και την ανεξαρτησία ενός οργάνου όπως η Όλαφ. Σε αυτά τα πέντε χρόνια εντολής που έχουμε στην Επιτροπή Εποπτείας, τι είδαμε, διαπιστώσαμε τις διάφορες δράσεις της Όλαφ οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή στην οργάνωση και στο σχεδιασμό των ερευνών. Κατά τρίτο, η Επιτροπή Εποπτείας από την αρχή της εντολής επέμεινε στην ανάγκη του να έχουμε ένα εγχειρίδιο, ένα σαφές εγχειρίδιο λειτουργικών ε, μεθόδων που θα αποτελούσε οδηγό για τους χρήστες σε όλη τη φάση της έρευνας. Το 2009 δημοσιεύθηκε η τελευταία έκδοση αυτού του εγχειριδίου και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία είναι βελτιώσιμα ε, κυρίως όσον αφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, διερευνουμένων ατόμων από την Όλαφ. Επίσης, ο ρόλος που, δίνουμε στην, ε, που προσδίδουμε στην Επιτροπή Εποπτείας μετά την απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου που επιτρέπει στην Επιτροπή Εποπτείας να έχει στα χέρια της προδικαστικές αποφάσεις που τις επιτρέπουν να βοηθήσει την Όλαφ στις έρευνές τους. Αυτή ήταν απόφαση, αυτό πλέον αποτελεί μέρος της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τώρα, στη φάση που βρισκόμαστε, Εμείς εργαζόμαστε για την μεταρρύθμιση του κανονισμού της ΟΛΑΦ, για τον κανονισμό 1073 και θέλουμε να συμπεριλαμβάνει πλευρές που θεωρούμε σημαντικές, που να μην έχουν μόνο σχέση με την πρακτική ή την ομολογία, αλλά να βρίσκονται στον τωρινό κανονισμό που θα προκύψει από τη μεταρρύθμιση του 1073. Θελήσαμε επίσης να υποβάλουμε μία πρακτική πρόταση και μία λιγότερη πρακτική πρόταση. Η έκθεσή μας δεν θέλει να είναι μελέτη ούτε θεωρητικός προβληματισμός. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν να μελετήσουμε έρευνες της Όλαφ από ε, έγγραφα και τεκμήρια ε, τα στοιχεία που εμείς ε, παίρνουμε στη μελέτη μας είναι πραγματικά στοιχεία Επίσης χρησιμοποιήσαμε και προηγούμενο υλικό, τις εννιάμινες εκθέσεις ε, και αξιολογώντας όλα αυτά τα στοιχεία αξιολογήσαμε τις τωρινές ρυθμίσεις το 1073 του 99, τον 285 του 96 την νομολογία του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και το πώς όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο εγχειρίδιο. Εμείς θέλουμε να υποβάλουμε προτάσεις, συστάσεις για την Όλαφ, για τον κάθε έναν από τους ε, ερευνητές τους, για τους μηματάρχες, για τους διευθυντές, τέλος πάντων για όλο το προσωπικό το οποίο εργάζεται στην Όλαφ και να ορίσουμε κριτήρια για την σχέση που μπορούμε να έχουμε μεταξύ Όλαφ και Επιτροπής Εποπτείας ούτως ώστε να πληρεί όλα τα στοιχεία τα οποία προανέφερα και αυτό στην επεξεργασία της ρυθμιστικής βάσης της Όλαφ. Εμείς ξεκινήσαμε από την ιδιάζουσα μορφή που έχει όλα. Πρόκειται για ένα διοικητικό όργανο ελέγχου, δεν έχει δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις. Όλες αυτές οι έρευνες περνάνε σε διάφορες φάσεις ε, ε, για να οριστεί το επίπεδο των ευθυνών, αν είναι διοικητικές ευθύνες, αν είναι ποινικές ευθύνες, αν χρειάζεται να ληφθούν μέτρα κλπ. Επίσης, διαφοροποιούμε και τις διάφορες έρευνες της ΟΛΑΦ, εσωτερικές έρευνες, εξωτερικές έρευνες. Η ΟΛΑΦ έχει διαφορετικές αρμοδιότητες στην κάθε μια από αυτές, όπως επίσης και στην χρήση εκ μέρους της Όλαφ των εσωτερικών διατάξεων των κρατών μελών. Διότι η Όλαφ ε, κάνει πολλές έρευνες, εσωτερικές έρευνες στα κράτη-μέλη και σέβεται τους ε, κανόνες ε, του κάθε κράτους μέλους για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τις προτάσεις τις χωρίζουμε σε δύο τμήματα. Πρόκειται για τις αναφορές για τις γενικές αρχές τις οποίες πρέπει να σέβεται η Όλαφ. Αντικειμενικότητα πρώτο, προσέχοντας τη σύγκρουση συμφερόντων. Δεύτερον, ανησυχίες όχι μόνο της ΕΡΟΛΑΦ αλλά και της Επιτροπής Προπολογισμών και των άλλων και της Κομισιόν κτλ. είναι το θέμα της καθυστέρησης η εργοπορία δηλαδή στις έρευνες και τελευταίο είναι η εμπιστευτικότητα των ερευνών της Όλαφ. Κάθε ερευνητικό όργανο θα πρέπει να σέβεται την, την ε, μυστικότητα γιατί αυτό αποτελεί το, τι θεμέλιο, το θεμέλιο λίθο. Είπαμε αντικειμενικότητα, διάρκεια, εμπιστευτικότητα. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που εγγυώνται την ανεξαρτησία της Όλαφ και των υποχρεώσεων της. Αφού λοιπόν ορίσαμε αυτά τα τρία ουσιαστικά στοιχεία, γίνεται και μία περιγραφή της διαδικασίας με όλες τις εγγύσεις που θα πρέπει να έχουμε κατά τις έρευνες της Όλαφ ε, στους διάφορους ε, τύπους ε, έρευνας, εσωτερικές ή εξωτερικές, αξιολόγηση, ξεκίνημα, άνοιγμα της έρευνας, ε, η έρευνα η ίδια, το κλείσιμο της έρευνας και το πώς όλα αυτά τα στοιχεία που προανέφερα γίνονται σεβαστά, δηλαδή πώς ανακρίνεται κάποιος, σε ποια γλώσσα, ε, τι πληροφόρηση πρέπει να δοθεί στον διερευνούμενο άτομο, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και είναι σημαντικό μία ειδική διάταξη η οποία θα επηρεάσει τις ε, έρευνες της Όλαφ ανάλογα με το τι έρευνα πρόκειται πρόκειται το προνόμιο και ασυλία της ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ε, τα προνόμια των υπαλλήλων ε, συνένεση που πρέπει ο Γενικός Γραμματέας ή ο Πρόεδρος ενός θεσμικού οργάνου να δώσει για να γίνει έρευνα ενός υπαλλήλου οι ειδικέ διατάξεις των κρατών μελών που θα πρέπει να είναι γνωστές να εφαρμόζονται πρέπει να ορίζονται μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ της Όλαφ και των διαφόρων οργανισμών ε, των κρατών μελών που κάνουν την ίδια δουλειά με την Όλαφ για να μην έχουμε παραβιάσεις ε, κατά τη διαδικασία. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προτείνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, ε, προτάσεις οι οποίες θα πάνε σε όλους τους ερευνητές της Όλαφ για να αξιολογούν σε κάθε στιγμή της έρευνας το πώς διαφυλάσσουν αυτά τα θεμελιώδη δικαίωμα. Και προοδευτικά θα αναθεωρούμε το λειτουργικό εγχειρίδιο για να ενσωματώνει αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις. και θα πρέπει να οριστεί ένα πραγματικό σύστημα ελέγχου της νομιμότητας των δράσεων της Όλαφ. Μόνιμος έλεγχος που πρέπει να ορίζεται ευθύ εξ αρχής. Και γι' αυτό πρέπει να ορίσουμε και να ενισχύσουμε τους εσωτερικούς μηχανισμούς της όλα για τον έλεγχο της νομιμότητας μέσα από τους τμήματάρχες, τους διευθύντες και όλη την γεραρχία για να καταλήξουμε στον Γενικό Διευθυντή. και μετά ειδικοί μηχανισμοί για τον έλεγχο της νομιμότητας, ας πούμε ειδικέ μονάδες που ήδη υφίστανται στην Όλαφ και που τα μέλη τους έχουν την, ε, νομική, την απαραίτητη νομική γνώση και ξέρουν πώς εκτιλήσονται διάφορες έρευνες. Οι ερευνητές επίσης θα πρέπει να καταρτίζονται για να αποφεύγονται τέτοιου είδους προβλήματα με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εγώ πιστεύω ότι με όλα αυτά που σας είπα, σας ανέφερα, τις ε, γενικές γραμμές αξιολόγησης αυτής της έκθεσης που είναι πολύ σημαντική, διότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, ε, τα υποστήριξε ούτως ώστε να μπουν στη συνθήκη της Λισαβόνας και αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε αυτή τη φάση έρευνα κλπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε που είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο εκπροσώπους της Επιτροπής Εποπτείας. Ευχαριστώ για και για τις γραπτές εκθέσεις που μας παρουσιάσετε προσωπικά. Ήταν πολύ πλήρης και εντυπωσιακέ. Μπορούμε να διαβάσουμε λοιπόν εντυπωσιακέ τοποθετήσεις στο θέμα αυτό που σας απασχολεί παραδείγματι την, τον έλεγχο νομιμότητας εντός της Όλαφ. Είναι θέματα που θα μας ε, απασχολήσουν φυσικά στη συζήτηση. Έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή Εποπτείας, μάλλον η έκθεση αυτή τη φορά είναι πολύ πιο έντονη στους όρους που χρησιμοποιούνται σε σχέση με προηγούμενες εκθέσεις. Έχω αναφερθώ στα εξή οκτώ σημεία. Καταρχάς ε, την προετοιμασία για την παρουσίαση από τον Επίτροπο των ε, προτάσεων του σήμερα το απόγευμα. Πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα τις ε, απαντήσεις και της Επιτροπής μας, αλλά αν έχετε κάποια ιδέα ήδη, γιατί η Επιτροπή Εποπτείας ήδη σε μεγάλο βαθμό έχει ενισχύσει τις εκθέσεις του Κοινοβουλίου. Και δεν βλέπω να ενισχύονται οι εξουσίες της ε, Όλαφ σε αυτό το κείμενο της Επιτροπής. Νομίζω ότι η πρόσβαση σε βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την Όλαφ. Και το θέμα αυτό ε, δυστυχώς δεν ρυθμίζεται στη νέα πρόταση του Επιτρόπου και έτσι δεν διευκολύνεται το έργο της Όλαφ. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι άποψη έχετε για το θέμα αυτό, τι πρέπει να κάνουμε. Δεύτερο σημείο. Στο χρονικό διάστημα αυτής τη έκθεσης έχουμε την χειρία τη θέση του Γενικού Διευθυντή και ε, μια γνωμοδότηση και για τον αναπληρωτή και βέβαια την στάση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, που ουσιαστικά ε, δεν έδρασε όπως θέλει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Επαγωπτίας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εάν έχετε κάποιες υποδείξεις, εάν διαπιστώνετε κάποιες ε, παρανομίες στην υπόθεση αυτή και εάν στις παρανομίες αυτές θεωρείτε ότι ε, στο βαθμό που μπορούσαν να προσαχθούν ε, ή να παραπεμφθούν οι υποθέσεις αυτά στα δικαστήρια, αν θεωρείτε ότι έγινε αυτό που έπρεπε να, να γίνει. Και επίση τώρα με τον κύριο Κέσλερ, Γενικό Διευθυντή πλέον και συγχαρητήρια για τη θέση του, ε, μεγάλο ποσοστό από ό,τι φαίνεται τον, του προσωπικού της, Ευρωπαϊκής της Όλαφ, με μετακύληση κατά 20% σε σχέση με τις προηγούμενες αναλογίες, τώρα ασχολείται μόνο με τις ανακρίσεις. Η εσωτερική λοιπόν αυτή μεταρρύθμιση της Όλαφ και η μετακύληση του προσωπικού πιστεύετε ότι έχει ολοκληρωθεί, χρειάζεται κάτι παραπάνω να γίνει. Και σε ποια σημεία θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να ε, επιληθούν τα προβλήματα με βάση τα όσα είχαν υποσχεθεί. Επίσης, ε, αναφέρεστε στην συντόμευση των διαδικασιών, ε, ιδιαίτερα σε ιστορικές διαδικασίες, πράγμα το οποίο χαιρετίζουμε. Ναι, αλλά όταν συντομεύουν έτσι διαδικασίες, μήπως τελικά δεν ε, διερευνώνται στον ίδιο αριθμό υποθέσεις. Μήπως δηλαδή γίνεται έρευνα λιγότερων υποθέσεων. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. με Στο έκτο μου σημείο, το de ως κανόνας, είναι δίκοπο μαχαίρι και είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου. Δεν ξέρουμε όταν ξεκινάμε αν πρόκειται για μια περίπτωση de minimis ή αν πίσω από αυτήν κρύβονται πολύ περισσότερα προβλήματα. Και νομίζω ότι η στρατηγική de minimis σημαίνει ουσιαστικά ότι η Όλαφ παρετείται από την εκδόταση κάποιων υποθέσεων, ενώ στην πραγματικότητα από πίσω τους κρύβονται πολύ χειρότερα σκάνδαλα. Και γι' αυτό θα ήθελα, με βάση και τον κανόνα de minimis, να μην δείξουμε πως ανεχόμαστε την ε, μικροεγκληματικότητα. Γιατί ήταν εσφαλμένο μήνυμα αυτό για την Ευρώπη και στη τελευταία ανάλυση δεν θα μας βοηθούσε καθόλου να καταπολεμήσουμε την πιο σοβαρή εγκληματικότητα. Ερωτώ λοιπόν, έχετε κάτι συγκεκριμένο σχέση με τον κανόνα de minimis, έχετε διαπιστώσει κάποια τέτοια παραδείγματα, πρέπει να γίνει μια ακρόαση ενδεχομένω. Στο έκτο σημείο που ανέφερε η κυρία Λόπε, εσωτερικέ και εξωτερικέ ε, έρευνες και αποκλίσεις μεταξύ αυτών. Εμείς θα θέλαμε να δούμε μια εξίσωση των δύο αυτών τύπων ερευνών ιστορικών και εξωτερικών, γιατί δεν θέλουμε το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει διαφορετική μεταχείριση από τη λυπή πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ρωτώ εσάς ποια είναι η θέση σα, γιατί θεωρείτε ότι θα πρέπει ενδεχομένω να έχουν διαφορετική και ευνοϊκότερη μεταχείριση οι υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι οι λοιποί πολίτε και με ποια διαδικασία θα πρέπει να γίνεται αυτό. Ε, στο 7ο σημείο λέτε στο 17ο, παράγραφο του εγγράφου σα ότι και πρόκειται για ένα σημείο το οποίο συζητούμε εδώ και χρόνια και πέρσι και πρόπερσι το συζητήσαμε ότι το εγχειρίδιο αυτό δεν έχει ακόμη προχωρήσει. Ε, το εγχειρίδιο της Όλαφ. Υπάρχει λοιπόν κάποια εξέλιξη. Μέχρι πότε πρέπει να περιμένουμε επιτέλους. Πότε μπορούμε να έχουμε κάποια σωστικά στοιχεία για αυτό το εγχειρίδιο. Και αυτά τα έστω μικροπροβλήματα θα τα ρυθμίσει το εγχειρίδιο νέου. Και στο 8ο μου σημείο, Βλέπουμε δύο εκπροσώπου τη Επιτροπή σα σήμερα. Όμω ο κύριο, και πολύ καλό είναι αυτό, αλλά ο κύριο Τρόμπερκ, κυριο στρομπερκ προεδρο τη Επιτροπή Εποπτεία έχει παραιτηθεί. Γιατί? ευχαριστώ. Ξεκινάει η συζήτηση. Ο συνάδελφος Μπάλτση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής Αποπτίας για την έκθεση την οποία συζητούμε. Θέλω να επενθυμίσω σε σχέση με την έκθεση αυτή ότι η Επιτροπή Εποπτείας συγκροτήθηκε για να ενισχύσει την ανεξαρτησία της όλο και για να βοηθήσει τον Γενικό Διευθυντή να επιτελεί καλύτερα τη δουλειά του. Η Επιτροπή αυτή, επομένως, συνεισφέρει τα μάλλα στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Όλαφ καθώς και στην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της Όλαφ. Η Επιτροπή αυτή παρακολουθεί, επιτηρεί σε διαρκή βάση δραστηριότητες της Όλαφ. Νομίζω ότι και η Επιτροπή αλλά και η εποπτική της δράση πρέπει να ενισχυθούν γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Όλαφ. Νομίζω ότι οι συστάσεις ε, που διατύπωσε η Επιτροπή είναι ορθές θα πρέπει να τις ε, υποστηρίξουμε, παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά την ποιότητα, τη διάρκεια των ερευνών. ή πτυχές οι οποίες έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τις προτεραιότητες, και επίσης σε σεβασμό των θεμελιωδών εγγύσεων σε σχέση με τις έρευνες πάντα, δημιουργία στρατηγικής, χάρη στρατηγική και πολλά άλλα ζητήματα. Να αναφέρω μεταξύ αυτών τις έρευνες οι οποίες είναι σε πρωτοκρατών μελών. Η κυρία Γκρέσλε ανέφερε κάποια σχετικά Ελπίζουμε η Επιτροπή αυτή να ενισχύσει την ποιότητα του έργου της Όλαφ. Θα μιλήσει και ο κύριος ε, Σεμέτα, ο Επίτροπος, ε, το μεσημέρι στην Επιτροπή μας. Ε, περιμένουμε κάποιες μεθοδολογικές πτυχές να μας σχολιάσει, να ακούσουμε κάποιες καινοτομίες και μετά από αυτή τη συζήτηση Νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι η αποτελεσματικότητα της όλα θα ενισχυθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η συνάδελφος Αγιάλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσοχή τους στα ζητήματα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο προσώπων όσο και ελεγχόμενων οργανισμών. Θα ήθελα να μου δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν τη διαδικαστική φάση στους ελέγχους στους οποίους προέβη η Όλαφ. Τώρα η εφαρμογή του περιφήμου εγχειριδίου το οποίο δεν πρέπει να είναι απλώς ένα εγχειρίδιο για πρακτικές οδηγίες αλλά θα έπρεπε να είναι και ένας ηθικός κώδικας και για τους διοικητικούς ελέγχους να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει κανένα ντεραπάζ, κανένα καμία παρασπονδία και πιστεύω ότι τον 21ο αιώνα μπορούμε να είμαστε ή ικανοί να αποφύγουμε τέτοιου είδους παρασπονδίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφές ε, ε, οντοτήτων ή μονάδων μετά από αυτούς τους ελέγχους. Πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε αυτά τα δικαιώματα και αυτές οι εγγύσεις να διασφαλίζονται. Και ρωτώ τον κύριο Λόπες, γιατί είναι αυτός ο οποίος ε, στάθηκε κυρίως σε αυτό το θέμα, για το θέμα των εγγύησεων τώρα που θα έχουμε ένα νέο διευθυντή στην όλα θα πρέπει να προχωρήσουμε και για τις συζητήσεις που έγιναν για την εκλογή του νέου διευθυντή ήθελα να ρωτήσω εάν είναι θετικό, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπα, ε, κάποιος ο οποίος έρχεται απ' έξω χωρίς να έχει μία προδικασμένη άποψη μπορεί να αποτελέσει και κίνητρο από τη μια αλλά και ε, συσπηρωτής και ενισχυτής από την άλλη για την ΟΛΑΘ. Ευχαριστώ η Κομισιόν, αν θέλει το λόγο. Δεν θέλει η Κομισιόν το λόγο. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή Εποπτείας, διότι η κυρία Γκλέσλερ αναφέρθηκε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην πρώτη παρατήρηση της κυρίας Γκρέσλε, αναθεωρημένη πρόταση μεταρρύθμισης, όπως είπα, κατά την ε, παρουσίαση της εκθεσής μας, δεν έχουμε μπορέσει ακόμη να το, να εξετάσουμε με το σύνολο του αναθεωρημένου κειμένου, θα το πράξουμε το χειτήριο δυνατό και στο βαθμό που μπορούμε θα συγκρίνουμε το ε, τι αλλάζει σχέση με το παρελθόν, τι θα έπρεπε να έχει αλλάξει και το καθεξής. Ε, μόλις λοιπόν λάβουμε το κείμενο θα ξεκινήσουμε μέσα στη δουλειά μας. Είναι προτεραιότητα και για μας. Στο, η δεύτερη παρατήρηση κυρίας Γκρέσλε δυστυχώς δεν αντελήφθη τι ακριβώς μας προτείνει. Σε, σε σχέση με την ε, ε, περίοδο κατά την οποία χείρευε η θέση του Γενικού Διευθυντή, είπατε ότι ενδεχομένω υπάρχουν παρανομίε και αν θα πρέπει αυτέ να παραμεθούν στα δικαστήρια. Αν έχετε κάποια στοιχεία, κυρία Γκρέσλε, γιατί εγώ δεν έχω υπόψη μου τίποτα τέτοιο. Για το 50% των απασχολουμένων τη Όλαφ που ασχολούνται με το ανακριτικό έργο είναι κάτι το οποίο εμεί ε, για χρόνια, για μεγάλο χρόνο μάλλον, προσπαθούσαμε να επιτύχουμε. Ευτυχώς ο κύριο Κέσλερ μας, δείχνει, μας λέει μας δηλώνει ότι ε, είναι ο στόχος που επιδιώκει και όπως λέει και η κυρία Γκρέσλε είναι πολύ ενθαρρυντική η, προ... η πρώτη τουλάχιστον εικόνα των σχεδίων και του προγράμματος του κυρίου Κέσλερ που μας παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα όταν τον συναντήσαμε και όπου μας παρουσίασε τις αδρές γραμμές της πολιτικής που θέλει να επιδιώξει. Βλέπουμε ότι είναι σύμφωνα με τα όσα εμείς εδώ και καιρό προτείνουμε. Επίσης η κυρία Γκρέστο σε σημείο 4 αναφέρεται στο κατά πόσον ε, η διάρκεια των ανακρίσεων είναι πιο σύντομη. Όντω, ερικές είναι πολύ πιο ε, τώρα οι δραστηριότητε ανάκριση και θα πρέπει να συγχαρούμε την ε, διεύθυνση Α που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ε, αν αυτό σημαίνει ότι εξετάζονται και λιγότερε υποθέσει, ναι, σε ένα βαθμό είναι λιγότερο ο αριθμό των υποθέσεων που εξετάζει η Όλαφ. Ε, επί παραδείγματι, γιατί έχω κάποια στοιχεία εδώ, 56 ανακρίσει είχε αναλάβει η διεύθυνση Α και 62 η Β, λιγότερε δηλαδή από την πρόπερση. Αυτά είναι τα περσινά στοιχεία. Άρα υπάρχει μια σχετική μείωση των υποθέσεων, ίσως όμως ήδη Όλαφ να έχει ε, λάβει υπόψη την επανειλημμένη σύστασή μας για προσδιορισμό προτεραιοτήτων των υποθέσεων με τι οποίε θα πρέπει να ασχολείται και έτσι φτάνω στην υπόθεση de minimis, μια πρόταση την οποία και εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε παρατηρήσει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις de ε, η Όλαφ δεν παρέλειψε να κάνει την έρευνα, την ανάκριση δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι δεν ε, ισχύει πάντοτε ο κανόνας de και ορισμένες φορές η Όλαφ όταν θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιοι όροι, υπόνοιες για ε, απόκρυψη σοβαρότερων εγκληματικών δραστηριοτήτων ε, δεν τον εφαρμόζεται ο κανόνα μήνυμης και πρέπει να πω ότι δεν έχουμε μεγαλύτερη ανοχή στα μικροεγκλήματα. Δεν είναι αυτός ο λόγος τον οποίο έχει εισαχθεί ο όρος δε μήνυμης. Άλλωστε από την προηγούμενη συνεδρίαση με την, ε, το Φεβρουάριο με την ε, με τον επικεφαλής της ΑΕΝΤΟΚ ε, συζητήσαμε το θέμα αυτό και υπόθηκε ότι θα πρέπει να ε, εξετάζονται και οι μικρότερες περιπτώσεις, λιγότερο σημαντικές αν θέλετε, μικρό μικροπαραβώσεις, μικροπαραβώσεις και τέτοια σε εσωτερικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο ούτε εγώ ούτε η όλα θα πρέπει να ανεχθούμε και οπωσδήποτε θα αντιμετωπιστούν εναρμόνιση εσωτερικών εξωτερικών ε, ανακριτικών ε, διαδικασιών θα το καλύψει ο κύριος Λόπες. Για το εγχειρίδιο, κυρία Γκρέσλε, έχετε δίκαιο. Είναι πολύ καιρό που απαιτούμε την ε, προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ζητούμε πολύ πιο συγκεκριμένους όρους και κανόνες που θα στηρίξουν όχι μόνο τις τη δουλειά των ανακριτών των ίδιων της Όλαφ, αλλά θα είναι χρήσιμο και ε, για την κοινή γνώμη, για τον δημόσιο χώρο, γιατί θα είναι βέβαια δημόσιο αυτό το εγχειρίδιο. Και θα ήθελα και η κυρία Αγία Σέντερ να μας πει τι θεωρεί ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει και ως κώδικα δεοντολογίας, όπως είπε ε, αυτό το εγχειρίδιο, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμη η σύσταση. Η τελευταία παρατήρηση της κυρίας Γκρέσλε την ε, παραίτηση του κυρίου Στρόμπερκ, του Προέδρου της Επιτροπής μας ολόκληρο το περσινό έτος και τους πρώτους, πρώτους τρεις μήνες, ο ίδιος μας είπε ότι ο φόρτος εργασίας που αντιμετωπίζει στη Σουηδία το, δεν του επιτρέπει να διατηρεί τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Αποπτίας. Γι' αυτόν τον λόγο φρονεί ότι δεν μπορεί ε, να επιτελεί τα διπλά αυτά καθήκοντα στο, στο επίπεδο ποιότητας που ε, επιθυμεί. Και ξέρετε ότι τώρα έχουμε την κυρία Τεάτο που όλοι, ε, που τη γνωρίζετε ε, και τη θυμάστε ασφαλώς ως πρόεδρο για το υπόλοιπο του έτους. Και τώρα μου επιτρέπετε ο κύριος Λόπες για να απαντήσει σε ερωτήσεις της κυρίας Γκρέσλε και της κυρίας Αγιάννα Σέντζερ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τη διαφορά των εσωτερικών και εξωτερικών ερευνών ή ανακρίσεων, ερώτημα της κυρίας Γκρέσλη και ότι θα μπορούσε να υπάρχει διακριτική μεταχείριση για, τους υποέρευνα, για τα υποέρευνα άτομα. Δηλαδή αν είναι υπάλληλοι, ανήκουν σε κάποιο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, να έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση από τους εκτός. Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα καλύτερης ή χειρότερης μεταχείρισης έχει να κάνει με τον ίδιο το χαρακτήρα των ερευνών, ε, που είναι διαφορετικές αναπερίπτωση, έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις, διαφορετικούς κανόνες και αυτοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και φυσικά πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης ε, όπως και σε οποιαδήποτε άλλο θεσμικό όργανο υπάρχουν κανόνες οι οποίοι είναι σε ισχύ και οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα οι έρευνες αυτές να είναι διαφορετικές αναπερίπτωση. Και σε κάποιες ε, περιπτώσεις η αντιμετώπιση τον μεν ή τον δε σε κάποια έρευνα, σε κάποια ανάκριση πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες. Αλλά επαναλαμβάνω ότι καταρχήν ε, ε, υπερτερεί και εφαρμόζεται πάντοτε η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης. Επαναλαμβάνω και επιμένω όμως ότι υπάρχουν οι κανόνες και θα πρέπει να τις ε, τηρεί τις διατάξεις αυτές κάθε ερευνητική, κάθε ανακριτική διαδικασία. Θα ήθελα να κάνω τώρα δύο σχόλια. Σε ό,τι αφορά την προθεσμία, κάτι το οποίο ανέφερε η κυρία Γκρέσλε, αλλά και η κυρία Γιάλα στην παρέμβασή της. Όπως είπα και στην αρχή, το ζήτημα της διάρκειας ε, των ερευνών, της ε, προθεσμίας, είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Η Επιτροπή μας ε, ευθύς εξ αρχής το είπαμε και το ξαναείπαμε και το ξαναμα τα είπαμε ότι πρέπει να διορθωθεί. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις διόρθωσης, μία μικρή άτολμη έτσι σιγανή βελτίωση τη βλέπουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει ξεκάθαρα να δούμε μέχρι πού πρέπει να φτάνει μια συγκεκριμένη φάση μια έρευνα. Και επίση θα πρέπει να υπάρχει ε, απαραίτητο υποχρεωτικά μια φάση αξιολόγηση, η οποία θα διαρκέσει την κατάλληλο χρονικό διάστημα για να δούμε τι έχουμε τι έχουμε στα χέρια μα. Σίγουρα δεν θα πρέπει να καθυστερούν για μήνε αυτέ οι διαδικασίε αξιολόγηση και μετά να λαμβάνεται η απόφαση για το κατά πόσο θα ανοίξει όχι. Θα ξεκινήσει όχι ανάκριση. Αυτό είναι σαφέ. και αυτό ε, πρέπει και λέγεται και στι διατάξεις ε, που ρυθμίζουν τη λειτουργία τη Όλαφ. Όπω έλεγα και στην αρχή, σε κάθε φάση τη διαδικασία ε, θα πρέπει να υπάρχει επιτήρηση και θα πρέπει να κρούμε τον κόδωνα όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ε, αδράνεια για μήνες σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Σίγουρα είναι κάποιες αποθέσεις δύσκολες ε, και χρειάζονται χρόνο, αλλά όταν βλέπουμε να μην υπάρχει καμία δραστηριότητα για μεγάλη χρονική περίοδο, αυτό πρέπει να προκαλεί να πυροδοτεί με έναν μηχανισμό, να υπάρχει έλεγχος και να βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται και να βλέπουμε τι κάνουν ε, και ο επικεφαλής μονάδας ε, και οι υπόλοιποι παιδιτές. πρέπει να παρακολουθούν ώστε να εξελίσσονται ομαλά οι διαδικασίες και να μην υπάρχει παράλυση όπως είπα. Τελευταίο σχόλιο για το εγχειρίδιο. Πράγματι το 2009 δημοσιεύτηκε η τελευταία έκδοση του εγχειριδίου η Επιτροπή είχε επιμείνει, είχε πει ότι είναι απαραίτητο. Παρά το ότι έχουμε μια βελτιωμένη έκδοση, διορθώνονται κάποιες λειτουργίες, βελτιώνονται κάποια πράγματα, το γεγονός είναι ότι κατά τη δική μας άποψη δεν είναι το κείμενο αυτό το οποίο χρειάζεται. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το κείμενο να είναι σαφές, να κάνει σαφή διάκριση των φάσεων και το κείμενο αυτό να μπορούν να, το, να μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές, οι οποίοι, τους ανακριτές οι οποίοι φτάνουν στην Όλαφ, να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως ένα μπούσουλα. Υπάρχουν διαφορετικοί φορείς, διαφορετικές ε, διοικήσεις στα 27 κράτη-μέλη, άλλη δομή και ο καθένας έχει τις δικές του ιδέες, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο εργασίας. Πρέπει πάντως να υπάρχουν κάποιες κοινέ γραμμές Έχουμε την ε, Ισπανική, Ιταλική, Σλοβακική αρχή ε, που έχουν τις δικές τους ε, διαδικασίες. Πρέπει κάπως να ομοιογενοποιηθούν. Όπως είπα, επιδέχεται βελτιώσει στο εγχειρίδιο. Προβλέπεται ότι μπορεί να τροποποιηθεί, άρα μπορούμε να το τροποποιήσουμε αυτό το εγχειρίδιο. Και αν είναι δυνατόν να τροποποιείται σε μόνιμη βάση, θα μπορούν να να, θα μπορεί να προσαρμόζεται με γνώμονα τις εξελίξεις που υπάρχουν αυτό το εγχειρίδιο. Δεν νομίζω υπήρχε και κάτι άλλο. Α, όχι, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, ο κύριος Γκάι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια συμπληρωματική ερώτηση προς την Επιτροπή Εποπτείας, ε, ύστερα από το άκουσα από τον κύριο Στρέμπερκ. Ε, για τον κύριο Στρέμπερκ, μάλλον. Είπατε ότι ε, παρετήθηκε πριν όμως οι φήμες που άκουσα εγώ έχουν να κάνουν μάλλον με υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του και το θέμα του διορισμού του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ. Υπέρβαση λοιπόν επί τη ευκαιρία του διορισμού. Παρακαλώ, θέλετε να απαντήσετε. Να σας πω. Ο λόγος που σας έδωσα ήταν ο λόγος που μας ανέφερε ο ίδιος ο κύριος Στρόμπερκ. Πολύ καλά, συνάδελφε Γκλέρ Γκρέσλερ, θέλετε να ανασύρετε τα συμπεράσματά σας. Ναι. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε από εδώ και μπρος, πώς συνεργαζόμαστε από εδώ και μπρος. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν, θερμά, να μας ετοιμάσετε μια γνωμοδότηση για την πρόταση της Επιτροπής με τις νέες προτάσεις για την περίοδο 2013 και μετά. Και θα ήθελα επίσης μια γνωμοδότηση προς το πώς βλέπετε την εσωτερική οργάνωση στην οποία θα πρέπει να κάτι τις μεταρρυθμίσει ο Γενικός Διευθυντής έτσι ώστε να απελευθερώσει από τα λοιπά καθηκοντά τους ε, αυτά τα ποσοστά, το 50% δηλαδή του προσωπικού που θα πρέπει να ασχοληθούν με τις ε, ανακριτικές εργασίες. Αυτά και πάλι βέβαια συμπληρωματικά των λοιπόν καθηκόντων της Επιτροπής σας που ευχαριστώ πολύ για τον πολύ καλό τρόπο που τις επιτελείτε. ήθελα λοιπόν να δω κάποια σχόλια για αυτή την τροποποιητική πρόταση, amending proposal, ώστε να δω τι γνώμη έχουν τα μέλη της Επιτροπής. Επίσης, δεν έχουμε δει, ιδιαίτερα όσον αφορά αυτή την αθεωρημένη πρόταση, συγκεκριμένα πώς θα λειτουργήσει, πώς θα εφαρμοστεί, ε, εάν δηλαδή σημαίνει και νέα εντολή εάν ε, από τον Νοέμβριο εφέτος υπάρξει νέα επιτροπή με νέα εντολή, πώς θα συνδυαστεί αυτή με την ενδεχόμενη επικάλυψη εργασιών και λειτουργιών της Επιτροπής Εποπτείας. Ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι. Κύριος Λόπες. Εγώ καταλαβαίνω και συμφωνώ με το ενδιαφέρον της κυρίας Γκρέσλερ η οποία πάντοτε ε, ε, θέλει, επιθυμούσε ιδιαίτερα το θέμα της ε, μεταρρύθμισης και ενίσχυσης του κανονισμού. Κοιτάξτε, η μεταρρύθμιση συνεχίζεται. Σε αυτά τα πέντε χρόνια ε, επεξεργαστήκαμε πολλές μεταρρυθμίσεις. Το κείμενο του 2008, το οποίο επεξεργάστηκε το Κοινοβούλιο, είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο. Μετά έγιναν και άλλες προτάσεις από την Κομισιόν. Και περιμένουμε κιόλας ήδη σήμερα το απόγευμα να δούμε ποια θα είναι η οριστική πρόταση. Εμείς εργαζόμαστε επ' αυτού, έχουμε επεξεργασμένα κείμενα τα οποία και τροποποιούμε όταν έχουμε κάτι το καινούργιο και έχουμε συγκριτικά κείμενα για τις θέσεις των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και όταν θα έχουμε την πληροφορία, τις πληροφορίες μας θα σας πούμε τη γνώμη μας αλλά όλα αυτά τα επεξεργαζόμαστε. Για την αναδιοργάνωση τώρα του γραφείου, εμείς έχουμε ένα νέο διευθυντή, Ήρθε όταν ανέλαβε ο άνθρωπος και μας μίλησε για την αναδιοργάνωση του γραφείου. Βέβαια μόλις ήρθε, μόλις έφτασε και πρέπει να ξέρει με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστεί, με ποιους θα αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες. για την οργάνωση της ε, ΟΛΑΦ και πιο συγκεκριμένα η κυρία Ράιτ ως εισηγήτρια εργαζόμαστε για αυτό το θέμα. Βλέπουμε για την τη συνεχή αναδιοργάνωση των τεσσάρων ε, ε, ετών η οποία Ε, η οποία έχει να κάνει και με το μάκρος, ε, με τη διάρκεια των ελέγχων, ας πούμε έλεγχοι που κρατάνε τέσσερα χρόνια είναι υπερβολική έλεγχη και πρέπει να διορθωθεί. Εμείς ε, είπαμε ότι για το Ιούνιο θα ολοκληρώσουμε τη γνωμοδότησή μας, θα αξιολογήσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις και θα κοιτάξουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς πρέπει να οργανωθεί το γραφείο για να λύσουμε προβλήματα που γνωρίζουμε ότι προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κι εσείς ή όχι. Θα ήθελα να πω ότι με ενθαρρύνει σπουδή με την οποία ο κύριος Κέσλερ ε, υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις του. Ξέρω ότι θέλει να προχωρήσει και να έχει το νέο σύστημα σε πλήρη λειτουργία μέχρι τις, ε, την επιστροφή από τις θερινές διακοπές, έτσι ώστε να ξεκινήσουν αυτές οι ανακριτικές διαδικασίες καινούριε από το φθινόπωρο. Θα κοιτάξουμε βεβαίως και τις νέες προτάσεις, ε, τις τελικές του προτάσεις δηλαδή, γιατί ξέρουμε ότι τώρα βρίσκεται σε επαφές με τα... με την εσωτερική ομάδα εργασία για τη διατύπωση αυτών των τελικών προτάσεων, έτσι ώστε να έχει έτοιμε τι ε, ιδέε αυτέ που οριστικοποιήσουν το έργο του. Είναι πολύ ενθαρρυντική λοιπόν αυτή η σπουδή. γιατί τη δική μα γνωμοδότηση, σχετική με την μεταρρύθμιση του 1073, θα την έχουμε μέχρι τον Ιούλιο φέτος. Ευχαριστούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης τη Εποπτεία συγγνώμη, της Όλαφ για αυτή τη σημαντική ακρόαση. Πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσια διάταξης για σήμερα το πρωί. Είναι η πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για τη Συνοχή και τη Στρατηγική σχετικά με την πολιτική της συνοχής και έχει το λόγο συνάδελφος Βόγκαν. Uh, Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση αυτή είναι για την Επιτροπή Περιφερειακή ε, ανάπτυξη, όχι την Επιτροπή ανάπτυξη, όπω λέγεται ε, στο έγγραφο. Βέβαια και η Επιτροπή Ανάπτυξη φαντάζομαι θα ενδιαφέρεται να το διαβάσει. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είμαι υπέρ των διαθροτικών ταμείων. Η πέμπτη έκθεση για τη συνοχή δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο και ήταν ε, μια άσκηση διαβουλεύσεων ε, που επακολούθησε μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Βέβαια το θέμα είναι αχανέστατο και την Επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξη ε, και περιλαμβάνει τις όλες τις ημερήσιες διατάξεις. Έχω λοιπόν συντάξει το σχέδιο γνωμοδότηση το οποίο απευθύνω σε όλου του συναδέλφου. Εκεί διατυπώνω κάποιε συστάσει. Πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχουν ένα περιθώριο σφάλματος 5% τα δεύτερα ταμεία, σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, παρόλα αυτά είναι βελτιωμένο το ποσοστό σε σχέση με το 11% της προηγούμενης χρονιάς και πολλά από τα σφάλματα οφείλονται στις πολύπλοκους κανόνες και διαδικασίες ε, που οι περιφέρειες, τα κράτη-μέλη και οι δικαιώσει σε τελική ανάλυση πρέπει να αντιμετωπίσουν. Οπότε και στις συστάσεις μου ζητώ απλούστευση των διαδικασιών η απλούστευση είναι μία λέξη που χρησιμοποιούμε κατά κόρον και πολλές φορές έχουμε συζητήσει τι θα πει απλούστευση, αλλά νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι να έχουμε συγκεκριμένες ιδέες για το τι σημαίνει απλούστευση για τον επόμενο γύρο ε, των διαφορετικών ταμείων. Έχουμε μιλήσει για τις πληρωμές, ότι οι πληρωμές ε, ε, ίσως θα πρέπει να ε, εφαρμόζουν ένα σύστημα κατά περισσότερο, να υπάρχει επίσης ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο θα συγκεντρώνονται διάφορα κονδύλια στο πλαίσιο κοινών διαδικασιών εφαρμογής. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις, οποίες δεν τυπώνω στην εκθεσή μου, μπορώ να τις διατρέξω γρήγορα-γρήγορα. Υποστηρίζω τις ε, δηλώσεις διαχείρισης ε, καθώς και την ανεξάρτητη γνωμοδότηση έλεγχου σε επίπεδο κρατών μελών γιατί έτσι θα ε, αυξηθεί η διοκτησία, η ιδιοποίηση εκ μέρου των κρατών μελών γιατί εκεί δαπανάται το μεγαλύτερο ποσοστό των κοντινών των ανθρωπικών ταμείων και επίσης τα κράτη-μέλη ε, καλό είναι να περάσουν από μια εθνική διαδικασία διαπίστευσης. Ε, έχουμε στη δική μου την ε, περιοχή, την Ουαλία κάνει κάτι αντίστοιχο, όπου η περιφερική κυβέρνηση και η Κομισιόν έχουν συνάψει μια, ένα συμβόλαιο αξιοπιστίας. Και βέβαια γίνονται έλεγχοι από την Επιτροπή, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών λόγω αυτού του συμβολέου αυτής της σύμβασης. Επίσης υποστηρίζω την αυτόματη διακοπή και αναστολή των πληρωμών όταν υπάρχουν ε, σοβαρές παρατυπίες και ελλείψεις. Βέβαια, τι θα πει σημαντικό, significant. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το ορίσουμε και ίσως πρέπει στην γνωμοδότηση να το συμπεριλάβουμε. Και τέλος, ε, στην ένατη σύστασή μου, λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος κυρώσεων που θα επιβαρύνει τα κράτη-μέλη και τους τελικούς δικαίους σε περίπτωση παρατυπιών. Ένα σημείο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι δεν θα ήθελα οι πληρωμές να συνδεθούν με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Κάποια κράτη-μέλη στηρίζουν τη διασύνδεση αυτή, αλλά νομίζω ότι θα ήταν τρέλα να απειλούμε ότι θα αφαιρέσουμε τα κονδύλια των ανθρωπικων ταμειων ταμείων από κράτη-μέλη και περιφέρειες που πλήττονται από οικονομικά προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό θα επιδεινώσει την κατάσταση, γι' αυτό δεν το συμπεριέλαβα στην εκθεσή μου. Επίσης, έχω συζητήσει με τον κύριο Σιγητή από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, τον κύριο Πίπερ, ο οποίο νομίζω ότι, ε, Πίπερ, ο οποίος νομίζω ότι συμφωνεί εν γέννη με τις συστάσεις μου. Και βέβαια αφού ακούσα τους συναδέλφους θα λάβω υπόψη μου ότι τυχόν έχουν να μου υποδείξουν. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Θέλει το ελεγκτικό συνέδριο. Η Κομισιόν. Η Κομισιόν θέλει το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. Από το κυρία Διευθύνση της Επασχόλησης και εκπροσωπώ και τις λοιπές γενικές διευθύνσεις που εμπλέκονται στην πρόσφαση. Με ενδιαφέρον καταγράφουμε τη γνωμοδότηση που πιστεύουμε καλύπτει κάποια από τα ερωτηματικά που μας απασχολούν και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν στην επερχόμενη μεταρρύθμιση. Επίσης, μεριζόμαστε τις ανησυχίε ε, που εκφράζονται ως με το Σαριάδη εμφανίζοντα ολόκληρη την έκθεση σε σχέση με την ε, παρατυπία ε, ή την νομιμότητα ορισμένων συναλλαγών αναφέρονται διάφορα κέρια ζητήματα ως προς τη διαχείριση και τον έλεγχο. Ολοκληρώθηκε τώρα η διαδικασία αυτή ανάλυσης των αποτελεσμάτων και συνεχίζουμε τις συνομιλίες ιδιαιτέρως με γνώμονες για να ολοκληρώσουμε τις προτάσεις που σκοπεύουμε να καταθέσουμε αυτό το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι και να αντιμετωπίσουμε βέβαια και τα προβλήματα που εντοπίζονται με την έκθεση. Είναι λοιπόν εν εξελίξει αυτές οι συζητήσεις και ως θεωρούμε ότι είναι πρόημο τώρα να ξεπεράσουμε στις δηλώσεις μας τα όσα περιλαμβάνονται στην πέμπτη έκθεση. Πριν όμως θα ήθελα να πω τα εξή. Ολίγα. Πρώτον, το συνεχιζόμενο έργο και τα θέματα που εγείρονται σχετίζονται και με τις εργασίες για τα διευθυντικά ταμεία και τους σχετικούς κανονισμούς, αλλά και με τους λοιπούς κανονισμούς. Το ζήτημα του ετήσιου κλεισίματος ε, λογαριασμών ε, με βάση και, τις, ε, και τη δήλωση αξιοπιστίας και τα όσα αναφέρει η γνωμοδότηση πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει σημαντικά το θέμα της αξιοπιστίας και ως εκ τούτου θα καλύψει πολλές από τις ανησυχίες που μας απασχολούν σήμερα και θα επιτρέψει να ε, καταγραφούν προτάσεις όπως αυτές που αναφέρει η Επιτροπή στο άρθρο 6, άρθρο 117 συγκεκριμένα της συνθήκης. 317. Για δε τις προτάσεις του κυρίου Βλεφτού, απλούστευση βεβαίως είναι στοιχείο κλειδί για τη βελτίωση της νομιμότητας και της ε, συμμόρφωσης των ε, διαδικασιών Αλλά βέβαια εδώ έχουμε και ένα ζήτημα με την απορρόφηση, άρα θέλουμε να κινηθούμε προς ένα σημείο, προς ένα σύστημα το οποίο θα μας, έχει, θα μας δίνει τη δυνατότητα να αμείβουμε για αποτελέσματα και όχι απλώς να δίνουμε δαπάνες, να πληρώνουμε δαπάνες, να εγγράφουμε μάλλον δαπάνες για εμπειρογνώμονες. Για τα θέματα που γύρονται στην τέταρτη, στην τέταρτο σύνολο προτάσεων που θα υποβάλει η Επιτροπή, σκοπεύουμε να τα απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφο Αγιάλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον Τέρεκ Βόγαμ ε, για τις ε, προτάσεις του και να ρωτήσω κι εγώ τόσο τον συνάδελφο όσο και την Κομισιόν. Πρώτο, για την Κομισιόν ρωτώ θα μπορούσε να μας δώσει αριθμητικά στοιχεία διότι εγώ ιστορικά πάντα το λέω δηλαδή αλλά κανένας δεν μου δίνει σημασία ούτε η Κομισιόν ούτε κανένας άλλος αλλά όταν μιλάμε εμείς για ποσοστά, εκατοστία ποσοστά ε, στην διαδικασία της δαπάνης και της εξπόστε και του εξπόστε ελέγχου των ε, δαπανών ε, για τα διαρθρωτικά ταμεία κλπ Το λάθος ε, στα λογιστικά τα βρίσκουμε μερικά χρόνια μετά. Και ρωτώ την ε, Κομισιόν. Οι τελευταίοι λογαριασμοί που φαίνεται να έχουν κλείσει οριστικώς είναι αυτές του 2000, 2000 έξι. Εμείς κλείσαμε οριστικά τους λογαριασμούς μέχρι το 1999 ή έχουμε κλείσει τους λογαριασμούς μέχρι το 2006. Και ρωτώ την Κομισιόν τι διαφορά έχει. Ας πούμε το 2005-2006 για παράδειγμα όταν διαπιστώνουμε το λάθος και, τον, και το τελικό κλείσιμο των λογαριασμών Ποιο είναι το ποσοστό λάθους. Εμείς με το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχουμε. Ας πούμε, ελέγχουμε τώρα το 2009. Με δύο χρόνια διαφορά. Και θα μας πούνε, το, το προβλέπω δηλαδή, το προβλέπω ότι θα έρθουν ε, τα λάθη και κυρίως όταν μιλάμε δηλαδή για, για, λάθη χοντρά τα οποία θα βγουν στον τύπο θα πούνε ορίστε τα λάθη που έγιναν στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι το ποσοστό λάθος ε, τα τελευταία 7 χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά. Αλλά φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από τη στιγμή που εμείς εγκρίνουμε τη διαχείριση μέχρι το κλείσιμο των λογαριασμών. Και δεν είναι τόσο το λάθος, ε, δεν είναι μόνο το χάσιμο των χρημάτων, δεν το έχουμε καταλάβει ποτέ αυτό. Και ρωτέτε το την Κομισιόν αν ποτέ θα καταφέρουμε όταν ελέγχουμε τους ε, λογαριασμούς ε, θα έχουμε και μία σειρά της διαδικασίας για το τι κάνουμε αλλά οι πολίτες πρέπει να ξέρουν την πραγματικότητα και όχι μόνο τους μεγάλους τίτλους της εφημερίδες, δηλαδή μόνο τίτλους για κρίσεις και κακά Και για τον συνάδελφο Βόγκαν ρωτώ, λέει στο σημείο 5 ότι είναι ικανοποιημένος με το νέο μέτρο το οποίο προτείνει η Κομισιόν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν μία έκθεση ανεξαρτήτου ελέγχου, ανεξαρτήτου audit. Και αυτή είναι μία φόρμουλα. Επίσης συμφωνώ με τον κύριο Βόγκαν όταν λέει ότι η Κομισιόν μπορεί να ζητάει από τα κράτη-μέλη να προχωρούν σε αυτούς τους ελέγχους αλλά τη βασική εποπτεία την έχει η Κομισιόν. διότι ναι μεν τα κράτη-μέλη πρέπει να δημιουργούν τα απαραίτητα όργανα για να ελέγχουν τη σωστή ε, να ελέγχουν τη δαπάνη και την ορθότητά της αλλά η Κομισιόν είναι σε τελευταία ανάλυση η υπόλογη που πρέπει να έχει την τελική εποπτεία και χαιρόμαστε γι' αυτό και για τις κυρώσεις ε, ρωτώ για ποιες κυρώσεις μιλάμε ο συνάδελφος Ντόιτς Ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι Όπω δείχνει άλλωστε η έκθεση, σκιώδη συγκητής για την πολιτική μου ομάδα είμαι εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σανφοβόν καταρχάς και να κεντρώθω σε τρία σημεία. Σύντομα σχόλια ουσιαστικά για την ε, συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να διαπιστώσω ότι ορθώς επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια σε θέματα πολιτικής συνοχής τα ποσοστά ήταν, όπως έδειχνε και η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, κάτω από το επίπεδο του 5%. και υπάρχει μάλιστα και μειωτική τάση. Αυτό έχει να κάνει όχι με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνο με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, η αποτελεσματικότητα των εργασιών μας θα πρέπει να ενισχυθεί, θα πρέπει ωστόσο και να αντιληφθούμε ότι το ποσοστό του σφάλματος υπάρχει με μειωτική τάση. Το 5% δηλαδή μειούται. ήθελα εδώ να εντοπίσω ένα σφάλμα ως προς τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει αυτό το ποσοστό σφάλματος στο ελεκτικό συνέδριο. Έχει δηλαδή το ελεκτικό συνέδριο το δικό τρόπο. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δικό της τρόπο υπολογισμού του σφάλματος και διαπιστώνω ότι οι δύο αυτές μέθοδοι ε, μεταξύ τους δεν ε, είναι ομοιόμορφες. Βλέπω απόκληση η οποία με ενοχλεί και ίσως επηρεάζει το επίπεδο του ποστοσφάλματος. Παράδειγμα από την Ουγγαρία, την πατρίδα μου. Η Βουδαπέστη είδε πολλές επενδύσεις από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στήριξη έγιναν οι έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα πόσο τομέα των δημοσίων, δημόσιας χρηματοδότησης 25% των επενδύσεων παρουσιάζουν ε, σφάλμα. 25% σφάλμα διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το ε, ίδιο αντικείμενο, το ελεκτικό συνέδριο διαπιστώνει το ίδιο ποσοστό το σφάλματος, αλλά καταλήξει το συμπέρασμα ότι συνολικά αυτές οι χρηματοδοτήσεις οδηγούν σε υψηλότερο ποσοστό σφάλματος. βρίσκει 100% δηλαδή σφάλμα το ελεγκτικό συνέδριο. Άρα δεν καταλαβαίνω, έχω ποσοστό 25% σφάλματος ή 100%. Είναι αυτό που λέμε, δεν γίνεται να είσαι ο λίγον έγκυος. Ή είσαι έγκυος ή δεν είσαι. Ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει. Ούτε ο λίγον ούτε πολύ. Αυτό μας λέτε με το 25% και το 100%. Λοιπόν, δεν είναι εδώ πέρα σωστή αυτή η διατύπωση και θα ήθελα να βελτιωθεί. Επίσης, θεωρώ πολύ σημαντικό να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου, πράγμα το οποίο ταυτόχρονα όμως σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να ζητήσουμε ριζική ε, μεταρρύθμιση των ε, θεσμών αυτών. Χρειάζεται μια απλούστευση φυσικά, ε, αλλά δεν αρκεί να την ζητάμε, πρέπει και να την εφαρμόσουμε. Για δε την εισαγωγή των κυρώσεων, για διακοπή των πληρωμών, ή άλλα μέτρα, εγώ θα ήμουν πιο προσεκτικός. Θα επέλεγα μια πιο διπλωματική διατύπωση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες λύσεις που να επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά ενός κράτους το οποίο έχει περιπέσει σε παρατυπίες, ενδεχομένω και παρανομίες σε σχέση με την εφαρμογή των κονδυλίων αυτών. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να προχωρούμε βήμα το βήμα. Και πιστεύω ότι με τις μεταρρυθμίσεις πρέπει να επιμείνουμε να εφαρμοστούν σωστά και όμως ταυτόχρονα φροντίζουμε να μην καίμε μαζί με τα, χλωρά, μαζί με τα ξερά και τα χλωρά έχουμε μια προσεκτική δηλαδή μεθοδολογία, χωρίς να λησμονούμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο χρειάζεται βέβαια βελτίωση, χρειάζεται μεταρρύθμιση, αλλά όχι και ε, διάλυση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το απορρίψουμε 100% για να εισαγάγουμε ένα νέο σύστημα. Ευχαριστώ κυρία Τσέσκοβα. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε όπως και άλλοι συνάδελφοι, καταλαβαίνω ότι η πολιτική συνοχής είναι πολύ επίκαιρη ως θέμα. Γνωρίζουμε ότι το 2013 θα είναι ένα έτος ε, μετέχμη για την πολιτική συνοχής εξού και μελέτησα το έγγραφο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης με ιδιαίτερη προσοχή. μελέτησα επίσης προσεκτικά και τη γνωμοδότηση του συναδέλφου από την Επιτροπή μας. Ένα πράγμα θέλω να τονίσω και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω λόγο γι' αυτό. Έχει αποτελέσει άλλωστε αντικείμενο πολλών συζητήσεων στην Επιτροπή μας. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει την ευθύνη για το ποσοστό σφάλματος σε ό,τι αφορά τους ε, σωστούς ελέγχους, ε, συμμόρφωσης προς τους κανόνες και σε ό,τι αφορά τις πληρωμές που γίνονται από το Ταμείο Συνοχής ή από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ποια είναι η ευθύνη των κρατών μελών, επίσης. Ποιο μερίδιο ευθύνη φέρουν τα κράτη-μέλη. Στα σημεία 5, 7 και 9 του σχεδίου γνωμοδότησης αναφέρονται σε αυτό και μιλούν και για κυρώσεις, οι οποίες θα πρέπει να επιβάλλονται και από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι στο μέλλον θα καταλήξουμε σε μια λύση που θα καλεί τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να είναι υπεύθυνοι για την επιβολή κυρώσεων. Θα ήθελα να έχω καλύτερη ενημέρωση για τις κυρώσεις, το είδος των κυρώσεων που προτείνουμε. Θα με ενδιαφέρει επίσης να δω κατά πόσο και πώς θα εφαρμόζονται, πώς θα επιβάλλονται οι κυρώσεις αυτές. η Κομισιόν, είτε με τι δικέ τη αρμοδιότητε, είτε μέσω των διαφόρων φορέων τη, θα μπορούσε να διενεργεί ελέγχου που τώρα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξή. Σε ποιο βαθμό αυτά που προτείνονται στην ε, γνωμοδότηση είναι ρεαλιστικά Πώς μπορούν οι φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης να διενεργούν ελέγχους ή να επιβάλλουν κυρώσεις στα κράτη-μέλη σε περίπτωση που η πολιτική συνοχής δεν εκτελείται σωστά. Αυτό είναι το σχόλιο που ήθελα να διατυπώσω και βέβαια περιλαμβάνει και κάποιες ερωτήσεις για τις οποίες θα ήθελα να ακούσω την απάντηση και μετά να αποφασίσουμε. Ευχαριστώ. Το ελεγχτικό συνέδριο θέλει το λόγο σχετικά. Παρακαλώ. Αξιότιμοι πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής αυτής. Ένα θέμα θέλω και εγώ να προσθέσω, γιατί νομίζω ότι οι υποδείξεις ε, που έγιναν, αλλά και η έκθεση του εισηγητή, αποτελούν ευτυχώς ένα πάρα πολύ, ε, μια πολύ καλή κατάληξη των πολλών προτάσεων που έχει διατυπώσει στην έκθεσή του τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Συνέδριο. Και σας ευχαριστώ γιατί έχετε συμπεριλάβει τις προτάσεις μας και έχετε ακολουθήσει τις συμβουλές μας. Θα ήθελα να προσθέσω ότι οι εννέα συστάσεις θα μπορούσαν να συμπληρωθούν λαμβάνοντας υπόψη την υπόδειξη την οποία έκανε ένας από τους ε, βουλευτές ε, της Επιτροπής, δηλαδή πώς θα πρέπει να ε, εκτελούνται οι διαγωνισμοί, πώς θα γίνεται η ανάθεση συμβάσεων. Γύρω στο 50% των σφαλμάτων, τα οποία εντοπίσαμε, είναι σφάλματα στον τομέα των διαδικασιών διαγωνισμού, στις προμήθειες, δημόσιες συμβάσεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Πρέπει όμως στο, διαγωνισμού διαγωνισμούς, στις δικασίες αυτές να υπάρξουν βελτιώσεις. Το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγή για το 2009, Είχε επίσης υπονοήσει ότι η Κομισιόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να εργαστούν στον τομέα της ποσοτικοποίησης των σφαλμάτων, στον τομέα αυτό, με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Διότι τα σφάλματα από τον τομέα αυτό τα ποσοτικοποιούμε με δύο μεθόδους. Να προσθέσω όμως αυτό δεν οδηγεί στην κατάσταση και είχα την εντύπωση ότι κάτι τέτοιο φεύγει να εννοηθεί, ότι τα ποσοστά σφάλματος έχουν προβληματική βάση. Δεν, δεν συμφώνω γι' αυτό. Θέλω να προσθέσω τα εξή. Το ποσοστό, τα ποσοστά σφάλματος μειώνονται τα τελευταία χρόνια. Το 2008 είχαμε γύρω στο 11% ποσοστό σφαλμάτων. 2009, στον τομέα αυτό πολιτικής, ήταν άνω του 5% το ποσοστό σφάλματος. Και να σας πω ότι εμείς κάνουμε διεξοδική ανάλυση, διεξοδικό έλεγχο του κάθε έτους, ξεχωριστά. Δεν είναι αυτόματο. Ούτε αναφέρεται ότι το ποσοστό σφάλματος ε, του 2009 στην προκειμένη περίπτωση που υπερβαίνει το 5% θα είναι μικρότερο από το 2009, από το έτος 2009-2010, θα είναι δηλαδή κάτω του 5. Μακάρι, μακάρι να είναι, το εύχομαι, γιατί αυτό θα δείξει ότι έχει βελτιωθεί η διαχείριση των ευρωπαϊκών οικονομικών και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Όμως, μπορεί να προκύψουν συνθήκες και καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε αύξηση αυτού του ποσοστού. Θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μια αυτόματη εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Από το 11 περίπου το 2008 στο 5 ή λίγο παραπάνω το 2000, ε, τα επόμενα χρόνια τέλος πάντων, 2009 και τα επόμενα έτη. Να προσθέσω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για το ότι οι υποδείξεις, οι συστάσεις σας ε, δείχνουν ότι οι δικές μας εκθέσεις, οι εκθέσεις του Λεπτικού Συνεδρίου αποτέλεσαν μια καλή βάση και ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια πιο χρηστή δημοσιονομική ε, διαχείριση του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε την Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα. να ρίξω μια να κάνουμε μια επισκόπηση των ε, ε, προτάσεων αυτών και θα με συμπληρώσουν, θα με διορθώσουν ενδεχομένω οι συνάδελφοι ε, για το θέμα του κλεισίματος των λογαριασμών. Αυτή τη στιγμή προχωρεί το κλείσιμο. Αν δεν απατώμε, έχουμε περίπου 20% των προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Υπάρχει μια μικρή απόκληση μεταξύ των ε, δύο κατηγοριών ταμείων και πληρώνουμε μόνο το 20% στο, στην αρχή του λειτουργικού προγράμματος. Στο τέλος δεν έχουμε το υπολογισμό του υπολείπου που στη συνέχεια μειώνεται κατά το ε, ανάλογο ποσοστό ε, επί της 100 εφόσον διαπιστωθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό σφάλματος. Άρα στο τέλος της περίοδου, αν είμαστε στο 100% ή λίγο, ή λίγο πάντων πιο μπροστά από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, μπορούμε να σας δώσουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για το ποσοστό σφάλματος, τι κίνδυνο έχουμε εντοπίσει, κίνδυνο σφάλματος δηλαδή, σε ποιο βαθμό μπορέσαμε να το ε, μειώσουμε με τις πληρωμές στα κράτη-μέλη. Άρα θα χρειαστούμε ακόμη μερικούς μήνες για να δώσουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Πάντως επισημάνατε και εσεί το θέμα των, ε, της που είναι και τα μεγάλα κενά. Όντως μπορεί αυτό να δίνει την εντύπωση ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εξού και συζητήσει ε, για τον δημοσιονομικό κανονισμό και τις αιτήσει σε καθάριση λογαριασμών. Αυτή είναι η διαδικασία ε, που μελετούμε αυτή τη στιγμή και ίσω να δείτε και να αντικατοπτρίσετε τι προτάσει τη Επιτροπής. Αργότερα και τα διορθωτικά ταμεία. Για τα όσα είπε ο κύριος Ντόιτς. Η μέθοδος που εφαρμόζει το Ελεκτικό Συμβούλιο ή η μέθοδος που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω τη διαφορά. Το Ελεκτικό Συνέδριο ε, στηρίζεται σε δείγμα ε, αριθμού λειτουργικού τοπικών παραγόντων ή ε, φορέων και συγκεκριμένου αριθμού κρατών μελών. Για να όμως επικεντρωθούμε σε ένα κράτος μέλος, δεν μπορούμε εμείς να χρησιμοποιούμε αυτό το, αυτό το ποσοστό. Χρειαζόμαστε ποσοστό σφάλματος για το κάθε κράτος μέλος. Επομένως δεν ξανακάνουμε ε, υπολογισμό εμείς, δεν διορθώνουμε δηλαδή τα αποτελέσματα, απλώς κάνουμε δικούς μας υπολογισμούς με βάση τα δεδομένα που μας προσφέρουν τα κράτη-μέλη. Simplification Uh, which you refer to uh, indeed action uh, Επίσης, απλούστευση είπατε. Η απλούστευση ναι, είναι πολύ σημαντική. Ε, έχοντας όμως εξετάσει και τελευταία μεταρρύθμιση του 1993 που πάλι είχε προβληθεί ένα της ε, απλούστευσης, δεν θέλω να επισημάνω ότι η απλούστευση καλή είναι, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά. Και αυτό και για λογαριασμό των δικαιούχων αλλά και ε, προς το ελεκτικό συνέδριο το μήνυμα σημαίνει ότι πρέπει η πραγματική απλούστευση να γίνει όταν ξέρουμε και που βρίσκονται, που εντοπίζονται τα σφάλματα. Στο κοινωνικό ταμείο έχουμε μικρή μικρότερους δικαιούχους, πολύ πιο περίπλοκο σύστημα, ενώ στο, στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι πιο συστημικά ενδεχομένω τα σφάλματα. Ε, αυτά. Εν νομίζω ότι έχουμε όμως μπει σε καλό δρόμο στην υπόθεση αυτή. Όσον αφορά τις κυρώσεις που ανέφερε η κυρία Τσέσκοβα. εξετάζουμε με τις δυνατότητες που έχουμε και τη δυνατότητα της διακοπής και της παρεμβάσεως και της άρσης των πληρωμών. Και αυτέ νομίζω ότι έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ποσοστού σφάλματο τα τελευταία χρόνια. Όπω αναφέρει και το Ελεκτικό Συνέδριο, από το 11% και μάλιστα πάμε και πιο παλιά, ακόμα υψηλότερο ποσοστό, στο τωρινό μα 5 περίπου αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το στοιχείο. Εντάξει, ναι, δεν αρκεί. Δεν αρκεί, αλλά είναι πάντως σημαντική βελτίωση. Και πάντως δείχνει ότι έχουμε πίσω στο σωστό δρόμο. Η Επιτροπή πάντως σκοπεύει να συνεχίσει τον δρόμο αυτόν και με τις αλλαγές που προβλέπουμε. Πιστεύουμε ότι θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Όπως πρέπει. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. για τα συμπεράσματα στον συνάδελφο Βόγαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τις παρεμβάσεις του. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την παρέμβασή του και για την ε, πρότασή του να συμπεριλάβουμε ένα δέκατο σημείο που θα αναφέρεται στι δημόσιε συμβάσει, στου διαγωνισμού. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για πολλά κράτη-μέλη, αλλά και για του δικαιούχου η διαδικασία, οι κανόνες ε, για τις προκηρύξεις, οι δεσμοπρατήσεις είναι πάρα πολύ πολύπλοκοι, οι κρατικές ενισχύσεις ε, και δεν ξέρω αν κάποιος καταλαβαίνει και αν καταλαβαίνει ας μας τα πει και σε εμά. Τώρα, στα σχόλια πάνω ε, για το ποσοστό σφάλματος ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου ανέφερε ότι από το 11 5% πέσαμε στο 5%, το είπε και ο κύριος Ντόιτς και έκανε και δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Δηλαδή ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να πέσει κάτω από το 5% το ποσοστό σφάλματος στο μέλλον. Και δεύτερον θα πρέπει να αναλάβουμε κάποιες δράσεις Ιδιότερα σε ό,τι αφορά την απλούστευση. Το είπα και εγώ στη δική μου παρέμβαση ότι μιλάμε πολύ για την απλούστευση αλλά χρειαζόμαστε πρακτικέ ιδέες για το πώ μπορούμε να απλουστεύσουμε τι διαδικασίε. και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε με τις περιφέρειες, με τους δικαιούχους, γιατί αυτοί είναι που συχνά παραπονούνται σε εμά για το πόσο πολύπλοκος είναι ο χαρακτήρας αυτών των διαδικασιών που ισχύουν. Θα πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν με τους δικαιούχους για να ακούσουμε και τις δικές τους ιδέες για το πώς μπορούμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Κυρία Τσέσκοβα και η κυρία Σέντερ επίσης έκαναν κάποια σχόλια. Και νομίζω ότι στο 5, ίσως και στο σημείο 6, αυτό το οποίο έλεγα εγώ από της ουσίας, ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις ε, διαχείρισης. Μόνο δύο κράτη-μέλη το έχουν εφαρμόσει, θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα και θα πρέπει οι δηλώσεις αυτές να υπογράφονται από τους υπουργούς. Να υπάρχει ένα είδος ιδιοκτησίας αυτών των δηλώσεων, αλλά και η Κομισιόν έχει ευθύνε. Έχει ευθύνε ό,τι αφορά τι δαπάνε των κοινοτικών κονδυλίων και νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβουν ε, και ε, οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευθύνη της και θα πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός που θα επιτρέψει την εξισορρόπηση αυτή. Έχουμε τις εθνικές δηλώσεις από τα κρατημέλη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ρόλο να διαδραματίσει. ολοκληρώνοντα να μιλήσω για τις κυρώσει γιατί κάποιοι συνάδελφοι το ανέφεραν. Η αναστολή των πληρωμών, η διακοπή των πληρωμών είναι, κάτι το προφανέ. Αλλά σε ό,τι αφορά επίση και την ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών είναι κάτι που ακούστηκε, είναι ίσως ε, μια ιδέα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, τα κρατημέλη μπορούν να ε, υποβάλουν τις τροπολογίες τους οι συνάδελφοι μέχρι την Παρασκευή. Θα λάβω υπόψη μου ό,τι είπε η Κομισιόν, ό,τι είπε το Ελληνικό Συνέδριο και ό,τι είπαν οι παριστάμενοι βουλευτές, αλλά σας καλώ να υποβάλλετε και γραπτές τροπολογίες μέχρι την Παρασκευή. Ευχαριστώ όλους σας, να τα πούμε στις τρει.